Καλησπέρα σας. Ε, ε, εκπλήσουμε που βλέπω μόνο δύο μέλη, αλλά σημαντικά. Οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι σήμερα αρχίζει η τρίτη εβδομάδα εργασιακής διαμάχης για τις επιβληθεί σε νέες συνθήκες εργασίας τους. Παρά τις πολλές παραχωρήσεις μας, η διοίκηση ουδόλως προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί μας για να λυθεί η διαφορά. Δυστυχώς σας πληροφορούμε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση ωραρίου και ότι η διερμηνία θα σταματήσει στις 6.30 ακριβώς. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Έχετε λάβει τα πρακτικά και την ημερήσια διάταξη. Αν δεν διαφωνεί κανεί, ε, εγκρίνουμε. Λεωνόρα, Εύη, συμφωνεί. Ωραία. Δεν έχω άλλε ανακοινώσει, ούτε διάφορα και θα περάσουμε αμέσω στο σημείο 5, που είναι η αναφορά 813 σχετικά μια ε, παραβίαση των κριτηρίων του τελικού καθεστώτος των ε, απορρίτων, ε, των απορρίτων <laughs> συγγνώμη, στην Ιταλία. Είναι εδώ οι αναφέροντες, οι δύο, για τέσσερα λεπτά, πέντε ο καθένας, θα σας ακούσουμε. Buongiorno e grazie. Καλημέρα σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Το ζήτημα τη αποτέφρωση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ιταλία και έχει να κάνει και με τα καύσιμα στερεά απόβλητα, που μόνο στην Ιταλία χρησιμοποιούνται και χαρακτηρίζονται ω καύσιμα, μολονότι είναι απόβλητα που δεν έχουν περάσει από διαλογή. Υπάρχουν πολλά ανησυχητικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με όσου ζουν κοντά σε τέτοιε εγκαταστάσει αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Στην Εμίλια Ρωμάνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αρμόδια αρχή παρακολούθηση καταγράφει πάρα πολλέ συνέπειε στην υγεία των πολιτών, ενώ φαίνεται ότι αυξάνονται οι περιπτώσει καρκίνου στο πάνκρεα, στο ύπαρ, στου πνεύμονε, στο εντερο σε οθήκε. Επίση εμφανίζονται πάρα πολλά κρούσματα λεμφώματο Χότκιν. Στο Τωρίνο τέθησε λειτουργία πρόσφατα μια μονάδα αποτέφρωση κοντά στην πόλη Γκέρμπιντο όπου βλέπουμε ότι οι οριακές τιμές που παράγονται εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ψηλές από αυτές οι οποίες προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε μια αύξηση 200% όσον αφορά τα στοιχεία αλουμινίου, αρσενικού, χρωμίου ή βαναδίου στα νύχια των μωρών. Όσοι ζουν στην κοιλάδα του πάγου επίση αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο στην έκθεση 13 2017 καταδεικνύει ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση ευθύνεται για 80.000 πρόωρου θανάτου στην Ιταλία. Με την επέκταση τη χρήση όμω των καυσίμων αυτών αυξάνονται και συνέπειε τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία των πολιτών και μάλιστα επιδεινώνονται. Αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, ιδίω για αυτού οι οποίοι ζουν πάρα πολύ κοντά σε τέτοιε εγκαταστάσει οι οποίε μολύνουν την ατμόσφαιρα. Λόγω της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης έχουμε χιλιάδες ή πολλές φορές εκατοντάδες χιλιάδες τόνους επικίνδυνων ουσιών που εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Επίση, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο στην Ιταλία τα εργοστάσια τσιμέντου βρίσκονται όλο και πιο κοντά στου οικισμού όπου κατοικούν πολίτε, όπω για παράδειγμα στην περιοχή Καλού Σκοτιντάντα, όπου κινδυνεύουν 20.000 πολίτε. Υπάρχει επίση μια πρόδουλη σύγκρουση ανάμεσα στα καύσιμα στερεά απόβλητα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά τα πλαστικά. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των καυσίμων αυτών το οποίο είναι πλαστικό και το οποίο δεν ανακυκλώνεται, χρησιμοποιείται ως πιο αποδοτικό απόβλητο παύλα καύσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτες με πολλά ανησυχητικά πορίσματα. Στην περιοχή Φάνα Εμανιάνγκο, μία μελέτη η οποία έγινε στην εκτροφή πουλερικών κατέδειξε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία πολυχρωμιωμένου δίφενηλίου στα πουλερικά τα οποία εκτρέφονται στην περιοχή αυτή, ακριβώ επειδή δίπλα υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγή τσιμέντου. Επίση, το ίδιο έχουμε δει και στην περιοχή Μονελίτσε, όπου από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να μετακινηθούν κάποια δημοτικά σχολεία, ακριβώ επειδή βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε τέτοιε μονάδε. Επίση, στην περιοχή του Αμπρούτσου φαίνεται από τι επίσημε περιφερειακέ αρχέ και τι εκθέσει του ότι οι επιπτώσει στην υγεία και στην ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνε για του πολίτε. Επομένω, βλέπουμε ότι οι μονάδε αποτέφρωση, καθώ επίση και οι μελέτε που έχουν έχουν γίνει για αυτούς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Αυτό λέγεται άλλωστε επίσημα και από το σχέδιο, από το πρόγραμμα ESCAPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και από το πρόγραμμα MAPEC Life Monitoring Air Pollution Effects on Children. Όλες αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις από τις εκπομπές των εργοστασίων τσιμέντου είναι πάρα πολύ επώδυνες για την υγεία των πολιτών. Και σαφώς θα πρέπει να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση περαιτέρω επέκταση των αποτευρωτών αυτών και των σχετικών εργοστασίων τσιμέντου. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μάρκο Καλντιρόλη. Okay. Σας ζητώ συγγνώμη. Τα εργοστάσια τσιμέντου σαφώ έχουν πάρα πολύ ε, δενέ επιπτώσει στο περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο πολλών ευρωπαϊκών νομοθεσιών, όπω για παράδειγμα των ρυθμίσεων που υπάρχουν για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν τεχνολογικά τα εργοστάσια αυτά. Βλέπουμε ότι ε, στα, ε, στα εργοστάσια αυτά τσιμέντου χρησιμοποιούνται ω καύσιμα διάφορα ρηκτά καύσιμα, τα οποία κλείουν στην ατμόσφαιρα πολύ σημαντικές ε, ποσότητες από ε, θείο. Επίσης πάρα πολλές ουσίες όπως για παράδειγμα διαλυτικά ή πολυχρωμένο ε, διφενήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, να καταφέρουμε να πετύχουμε μία μείωση των οξύδων του αζότου και του οξύδου του θείου που εκπέμπουν τα εργοστάσια αυτά. Και δυστυχώ η Ιταλία είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ενέκρινε μία εθνική νομοθεσία η οποία αναγνωρίζει τα αποχαρακτηρισμένα απόβλητα ω απόβλητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καύση στα εργοστάσια παραγωγή τσιμέντου. Βλέ Βλέπουμε, γνωρίζουμε μάλλον ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμα και στη Γερμανία, χρησιμοποιούνται απόβλητα ω καύσιμα στα εργοστάσια παραγωγή τσιμέντου, αλλά στι χώρε αυτέ, όπω τη Γερμανία, εξακολουθούν και χαρακτηρίζονται ω απόβλητα. Ανταυτού βλέπουμε ότι στην Ιταλία παρακάμπτεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρησιμοποιείται μια άλλη διαδικασία αδειοδότησης και τα καύσιμα αυτά χρησιμοποιούνται ως αποχαρακτηρισμένα πλέον απόβλητα, ως end of waste, όπως λέγεται στα αγγλικά. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν γίνονται οι απαραίτητε μελέτε περιβαλλοντικού αντικτύπου και ούτε μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι πολίτε στι μελέτε αυτέ όπω προβλέπεται από την Οδηγία 75 του 2016 τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι εκπομπέ, όπω για παράδειγμα ταξίδι του αζότου, με διαφορετικού τρόπου. Με τεχνικέ δηλαδή παρεμβάσει στη μονάδα παραγωγή και με νέα συστήματα επεξεργασία των εκπομπών. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ιταλία βασίζονται σε κάποιε επιδοτούμενε μελέτε για να αποδείξουν τελικά ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τα απόβλητα αυτά ω καύσιμα, τα λεγόμενα αποχαρακτηρισμένα απόβλητα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι στι μελέτε αυτέ καλύπτονται πολλά ετερογενή εργοστάσια που έχουν εντελώ διαφορετικέ εκπομπέ και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πολύ κατώτερο του πραγματικού. Μόνο αν γινόντουσαν εντελεχεί μελέτε και αναλύσει και συγκεκριμένα εργοστάσια θα βλέπαμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το τσιμέντο το οποίο παράγεται κατά αυτόν τον τρόπο, η πρόεδρο διακόπτη, δεν μπορείτε να συνεχίσετε. 5 ε, λεπτά είχατε στη θέση, έχετε καταναλώσει ήδη τα 6 λεπτά. Αφού πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω μπορεί να ξαναπάρετε το λόγο αν θέλετε για να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σα. Θα πρέπει τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει ακόμα γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι δεν είναι. Επομένω, προσμένουμε την προφορική σα τώρα απάντηση. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρούσα ότι είχατε λάβει τη γραπτή μας απάντηση, ίσως ακόμα να την προετοιμάζουν οι υπηρεσίες μας, τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω προφορικά να απαντήσω. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ που μας επισημαίνουν αναφέροντες είναι η χρήση αυτών των απορριμμάτων ως σε καύση σε ορισμένα στις ορισμένε εγκαταστάσεις. Εφαρμόσαμε τα κριτήρια της οδηγίας ε, πλαίσιο και συγκεκριμένα του άρθρου 6 για τα απόβλητα. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν, δεν έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση κριτήρια, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν τα δικά του. Αυτό έπρεξε η Ιταλία και έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό περί τεχνικών μέτρων. Ε, αυτό είναι μια αρχική εγγύηση που εγγυάται την αντικειμενικότητα των κριτηρίων και ότι λαμβάνουν υπόψη τους την νομοθεσία για το περιβάλλον. Ωστόσο, εφαρμόζεται επίσης και η οδηγία για τις εκπομπές των εργοστάσεων και ε, από αυτήν προκύπτει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες δυνατές τεχνικές ε, λύσεις που μπορούν να αγγιηθούν την προστασία του περιβάλλοντος. Και οι δύο αυτές οδηγίες στόχο έχουν να προστατεύσουν το περιβάλλον στο ύψιστο δυνατό επίπεδο με βάση τα επιστημονικά δεδομένα σε αυτήν την περίπτωση που συζητούμε δεν υπάρχουν στοιχεία ε, που να αποδεικνύουν ότι έχουν παραβιαστεί οι δύο αυτές οδηγίες όσον αφορά την ε, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο δεν ακολουθεί αυτές τις διατάξεις, τότε οι εθνικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν δράση, δηλαδή να εξετάσουν κατά πόσον υπάρχει μια τέτοια παράβαση και αν ναι, να, να, να, να ε, ασκήσουν την απαιτούμενη δίωξη, να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει. Δεν είναι αυτό μια αρμοδιότητα της Επιτροπής, αλλά των εθνικών αρχών. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η νομοθεσία Ιταλική συνάδει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντικο. Κυρία Εύη έχει το λόγο και τα υπόλοιπα μέλη συνεχεία. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά την απάντηση που μόλις τώρα μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, οι αναφέροντε δεν αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, σε ένα συγκεκριμένο δηλαδή εργοστάσιο, αλλά σε ένα συστημικό πλέον πρόβλημα που εμφανίζεται στην Ιταλία όσον αφορά τις εθνικές νομοθεσίες. Και προφανώ αναφέρομαι στο διάταγμα κλίνη του 2013, όπου προβλέπεται αυτός ο αποχαρακτηρισμός των αποβλήτων και που ουσιαστικά το διάταγμα αυτό δημιούργησε μια τεράστια αγορά για τη χρησιμοποίηση των στερεών αυτών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα όχι μόνο ιταλικό αλλά και ευρωπαϊκό. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο βασίζεται ακόμα στην χρήση της αποτέφρωσης ως βασικός μηχανισμός, ως βασική μέθοδος για την επεξεργασία των αποβλήτων. Για ποιο λόγο το λέω τώρα αυτό. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δευτερεύον κάψιμο στέρεο απόβλητο και να χρησιμοποιηθεί εν συνεχεία σε μια βιομηχανία που παράγει για παράδειγμα τσιμέντο, δημιουργείται παράλληλα μια τεράστια αγορά επεξεργασίας του αποβλήτου αυτού, το οποίο δεν σταματάει πλέον να θεωρείται απόβλητο και γίνεται καύσιμο και καταλαβαίνετε ότι αυτό βάλει κατά τη ίδια τη αρχή της κυκλικής οικονομία που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προωθεί η ίδια η Ευρώπη. Ξέρετε ότι πάρα πολλέ φορέ αντιμετωπίζοντα πάρα πολλέ δυσκολίε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πλήρω τι αρχέ τη κυκλική οικονομία. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια σαφή θεωρώ κατάσταση με πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά τη χρήση αυτών των CCS, των καύσιμων στερών αποβλήτων, και βλέπουμε ότι δημιουργούνται επιπτώσεις όχι μόνο σε επίπεδο ανθρωπινής υγείας, καθότι ε, καίγονται στα εργοστάσια τσιμέντου τα προϊόντα αυτά και ξέρετε ότι τα εργοστά αυτά, αυτά τσιμένου έχουν ε, κλιβάνους οι οποίοι όμως είναι για την καύση άλλων προϊόντων, άλλων καυσίμων και όχι για την καύση αποβλήτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για την καύση ενός πολύ επικίνδυνου προϊόντος, ενός προϊόντος που δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να θεωρείται καύσιμο, αλλά που παραμένει ένα απόβλητο. Τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία παρήγαγαν, όπως γνωρίζουμε, μονοξίδιο του αζότου, θα μπορούσαν τουλάχιστον να περάσουν από μια διαδικασία που θα οδηγούσε σε μείωση αυτών των εκπομπών. Ανταυτού όμως το μονοξίδιο του αζότου πάβει πλέον να είναι πρόβλημα. Δεν έχουμε τόσε πολλέ επικίνδυνες εκπομπέ μονοξίδιου του αζότου, αλλά έχουμε πλέον πολύ πιο επικίνδυνα στοιχεία, τα οποία περιέχουν βαρέα μέταλλα, πολλέ φορέ διοξίνε και κατά αυτόν τον τρόπο απειλείται ακόμα περισσότερο τελικά η υγεία των πολιτών. Το αίτημά μας λοιπόν είναι προφανώς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή προκειμένου να μπορέσουμε και στο μέλλον να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ ε, πώ διαμορφώνεται η κατάσταση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ζητάμε επίση ε, να γίνει μια ανακοίνωση σε εθνικό επίπεδο, μια γνωστοποίηση τουλάχιστον προς το, περιβάλλον, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ιταλίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αγώνας αυτός που η μάχη αυτή που πραγματικά καταβάλουμε ως κίνημα των πέντε αστέρων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζητάμε λοιπόν ότι θα πρέπει αν μη τι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει ένα χειρό μήνυμα προκειμένου να λάβει έγκαιρη δράση η Ιταλική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει επίση να γίνει και μία ενδελεχή μελέτη, προκειμένου πραγματικά να καταφέρουμε να δούμε όλου του αστάθμητου παράγοντε όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Α μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή τσιμέντου ενέχει πάρα πολλά κατάλοιπα εν συνεχεία, τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και για το ζήτημα αυτό να αρχίσουμε να διεξάγουμε διάφορες μελέτες, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ε, θέτουμε κινδύνο, σε πάρα πολύ σοβαρό κίνδυνο, την ίδια την υγεία των πολιτών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πιεντιτσίνη. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, εξ ονόματο του κινήματο των Πέντε Αστέρων και πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσα να σα παρουσιάσω την δική μου την εμπειρία από τι εργασίε που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή περιβάλλοντο και οι οποίε θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε και για την Επιτροπή Αναφορών. Θεωρώ όμω ότι η γνώση αυτή θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και για του ίδιου αναφέροντε, καθότι αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιο καιρό, στην Ιταλία έχουμε αρχίσει να ασχολούμεθα πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό και το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει προφανώς και στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για διοξίνε, για αλουμίνιο, για βαρέα μέταλλα, για όλα αυτά τα οποία εκλείονται από την παραγωγή τσιμέντου ή τσιμέντου τύπου κλίνκερ από τις ε, από τις μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Θα ήθελα παρόλα αυτά να επιμείνω σε αυτά τα οποία κάνουμε επιτόπου. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε διάφορες παρουσιάσεις σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας όπου βρίσκονται μονάδες παραγωγής τσιμέντου που χρησιμοποιούν τεχνικές αποτέφρωσης, ιδίως τεχνικές αποτέφρωσης για κάψιμα στερεά απόβλητα. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν, όπως σας είπα, διάφορες δράσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται αυτά τα εργοστάσια. Σε, σε μια πρώτη φάση λέμε ότι το σχετικό διάταγμα του Φεβρουαρίου του 2013 της Ιταλίας ουσιαστικά αποχαρακτηρίζει διάφορα απόβλητα τα οποία θα έπρεπε να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται απόβλητα. Επίσης η οδηγία του 2008, 98 του 2008, της 10ης Νοεμβρίου του 2008, λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και ότι δεν μπορούν τόσο εύκολα να να... ορισμένα απόβλητα να θεωρείται ότι πάβουν να αποτελούν απόβλητα αν έχουν υποστεί, υποστεί εργασία ανάκτηση κτλ. Γιατί ακριβώ πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνα. Έπειτα, η οδηγία του 2006 που είναι υπεύθυνη για την καταγραφή, τη χρησιμοποίηση και την απόσυρση των χημικών ουσιών, η οδηγία ουσιαστικά REACH, θα πρέπει να ισχύει και για το τσιμέντο Clinker. Μόνο αν το τσιμέντο αυτό ουσιαστικά περιέχει φυσικά στοιχεία, όχι στοιχεία τα οποία έχουν προέλθει από χημική επεξεργασία. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως το τσιμέντο τύπου κλίνκερ είναι ότι πραγματικά είναι ένα τσιμέντο το οποίο απορρέει από χημικές επεξεργασίες και όχι από στοιχεία τα οποία βρίσκονται φυσικά στο περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα καύσιμα στερεά απόβλητα περιέχουν βαρά μέταλλα καθώς επίσης και αλουμίνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία θα μπορούσα μάλιστα να δώσω όλες αυτές τις πληροφορίες τους αναφέροντες, πληροφορίες τις οποίες έχουμε συλλέξει σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Ανάλογες δράσεις και ενημερώσεις θα γίνουν επίσης και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας όπου βρίσκονται αποτεφρωτές και μονάδες παραγωγής τσιμέντου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχουν πάλι αναφέροντες για άλλα δύο λεπτά και δεχομένω, κύριε Καλτιρόλη να συνεχίσετε και την παρέμβασή σας από το σημείο που σας διέκοψα τόσο απότομα πριν από λίγο. Θα μπορούσατε πάντως να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε όλο το κείμενό σας, γιατί το έχουμε ήδη λάβει. Ενδεχομένω θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ανταποκριθείτε στα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνάδελφοι της Επιτροπής. Και εν συνεχεία θα προσπαθήσω εγώ να συνοψίσω την όλη συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Ένα ζήτημα θα ήθελα να θίξω μόνο, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της μας είπε ότι η εθνική νομοθεσία, η ιταλική δηλαδή νομοθεσία, εν προκειμένου, όντως ε, καταδεικνύει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ένομα, σύνομα ουσιαστικά τα καύσιμα αυτά, τα απόβλητα αυτά ως καύσιμα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχει γίνει και μία πρώτερη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανταποκριθεί λέγοντα ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την αρνητική χρήση των ε, αποβλήτων αυτών. Παρ' όλα αυτά όμω ούτε τα αντίθετα στοιχεία υπάρχουν, δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα μελέτε, οι οποίε εμπεριστατωμένα να λένε ότι όντω δεν υφίστανται βλαβερέ συνέπειε από τι εκπομπέ αυτέ για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία. Και όπως πολύ σωστά είπε ο προλαλής σας, ο Ευρωβουλευτής, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιληφθεί του ζητήματος αυτού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, να εκπονήσει δηλαδή μία ενδελεχή μελέτη και να εξετάσει λίγο περισσότερο την παραγωγή τσιμέντου στα πλαίσια της οδηγίας REACH. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε πλέον το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ας προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε. Βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να περιμένουμε και τη γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε πλήρως όλα τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνετε αλλά φυσικά χρειάζεται να τα δούμε και γραπτός όλα αυτά για να τα μελετήσουμε ενδελεχώς. Θα πρότεινα λοιπόν τώρα να το κάνουμε, να αναλύσουμε την γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να στείλω και επιστολή στην Ιταλική κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ ενισχυτικά όλα αυτά και ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών έχουμε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και ανησυχούμε και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι θα ήταν ε, χρήσιμο κάτι τέτοιο. Συμφωνούμε από αυτού. Ωραία. Καλώς. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν. Και βλέπω να χαμογελούν οι αναφέροντες, πράγμα που δεν συμβαίνει και συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να ε, τονίσετε και να μας επισημάνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και καλό σας απόγευμα στις Βρυξέλλες, ακόμα και αν ο καιρός δεν είναι τόσο καλός όσο στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, όσο είστε εδώ, προσπαθήστε να χαρείτε τις Βρυξέλλες. Και ε, πάμε στην επόμενη αναφορά 595 σχετικά με την αντλητική υδροελεκτρική εγκατάσταση σάλας Ασκόνσας στην περιοχή Ορένζε. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, δεν έχω πια βουλευτές. Ήθελα να σας επιστήσω την κατάσταση ε, των διερμηνέων και περίμενα για να δώσω το λόγο στους ε, διερμηνείς όταν θα έρχουν πολλοί βουλευτές οι περισσότεροι. Δεν ξέρω, θέλουν τώρα να κάνουν την ανακοίνωσή τους οι διερμηνείς. So, I give you some 30 seconds. Σας δίνω 30 δεύτερα. Οι διερμηνείς σα ενημερώνουν ότι σήμερα αρχίζει η τρίτη εβδομάδα εργασιακή διαμάχη για τις μονομερώς επιβληθήσεις νέε συνθήκε εργασία του. Παρά τις πολλές παραχωρήσεις μας, η διοίκηση ουδόλω προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί μα για να λυθεί η διαφορά. Δυστυχώ σα πληροφορούμε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση ωραρίου και ότι η διερμηνία θα σταματήσει στις 6.30 ακριβώ. Σα ευχαριστούμε για την προσοχή σα. Thank Ευχαριστώ πολύ είναι όλοι εγνώση ε, του γεγονότος ότι θα πρέπει να τηρούμε το ωράριό μας και σήμερα ακόμα περισσότερο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη αναφορά. Ο αναφέρον απουσιάζει, αλλά πάντα παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και έχει το λόγο. Η κυρία Μελίν Βάργα θα πάρει το λόγο ή κάποιος άλλος ή ο κύριος Καβαδάς. Ελίσσα Βάργα Αμελίν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Εφόσον απουσιάζει ο αναφέρον, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα και στο περιεχόμενο της λόγω αναφοράς. Ε, ο αναφερόμενος παρουσίασε την κατάσταση. Είναι μια υδροηλεκτρική εγκατάσταση ε, για την ε, άντληση υδάτων μεταξύ δύο ταμιευτήρων. Ο ένας ταμιευτήρας είναι στη Σάλας που είναι σε προστατευόμενη περιοχή και το νερό είναι καλής ποιότητας. Ο άλλος ταμιευτήρας βρίσκεται στην περιοχή Κόντσας που δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση και λέει ο αναφέρον ότι κινδυνεύει να μολυνθεί το νερό ε, στην Σάλας όπου τα μυευτήρα είναι καλύτερη ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο έστειλε απάντηση, ωστόσο θα ήθελα να τονίσω ότι ζήτησε επιπλέον ενημέρωση την περασμένη Παρασκευή 15 έκτου 2018 αναφέρον και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη αυτή την επιπλέον πληροφόρηση. Καταρχάς Θέλουμε να θυμίσουμε ότι το κράτο μέλο είναι αρμόδιο προκειμένου η Ισπανία για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών ε, και τα περιβαλλοντικά. Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, έχουν γίνει τα βήματα που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου επιπτώσεων. Έχει γίνει δημόσια διαβούλευση και επίσης ε, δημοσιεύτηκε η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Στη διαδικασία αυτή έχουν εντοπιστεί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι αλλά και τα δυνατά μέτρα πρόληψης των κίνδυνων αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η έγκριση ή η η διαδιοδοτηση του έργου δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί από την αρμόδια αρχή που εμπροκειμένο είναι η Ιδρογραφική Συνομοσπονδία του Μίνιο Σιλ. Τονίζω, το έργο ακόμα δεν έχει λάβει έγκριση για να εκτελεστεί. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για μια διοικητική πράξη ε, κατά της οποίας μπορεί κανείς να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων ισπανικών αρχών. Σε ό,τι αφορά τις επιπλέον πληροφορίες που έλαβε ο αναφέρον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι και πάλι τονίζουν τον κίνδυνο ή τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με το έργο και τονίζουν την κατάσταση των υδάτων στην περιοχή. Ιδιαίτερα αναφέρονται σε μια σειρά από υδάτα που δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι το υδρολογικό σχέδιο του Μουνιοσίλ προβλέπει διάφορες εξαιρέσεις Οπότε, η διεύρυνση της προθεσμίας ε, για τους περιβαλλοντικούς στόχους προβλέπεται. Δηλαδή, υπάρχουν τεχνικά μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των υδάτων. Λοιπόν, για να ολοκληρώνω, με την πληροφόρηση που έχουμε αυτή ε, τη στιγμή στη διάθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι το έργο αυτό μπορεί να παραβιάσει τις οδηγίες που αναφέρει ε, στην αναφορά του ενδιαφερόμενος. Ε, αυτά, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω είναι εύκολο να συνοψίσουμε. Μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν διαπιστώνει να υπάρχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις από πλευράς Natura 2000, ε, παρά το γεγονό ότι ο υδροφόρος ορίζοντας επηρεάζεται. Όμως, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια αλλά κατά τα άλλα από τη δική μας την πλευρά θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά γιατί διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κάποια παραβίαση όσον αφορά το Natura 2000 ή την νομοθεσία την περιβαλλοντική. Μια, από τα δύο μέλη που είναι παρόντα ρωτώ, συμφωνείτε, ναι. Θέλετε το λόγο, όχι. Μόνο γιατί μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα είπε η Πρόεδρος, να κλείσει η αναφορά και απλώ να το παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, Ιγκόρ, είμαστε τρεις και συμφωνούμε και οι τρεις ομόφωνα. Τέλεια, φανταστικά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Δεν περιμένουμε αναφέροντα εδώ. Είναι η 614 σχετικά με τη σύνδεση του οικοπαίδου του αναφέροντος στο δημόσιο δίκτυο ίδρυυσης. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε μια κυρία που έχει, ε, περίεργο όνομα και δύσκολο, ο Τζαράμπαλ Φερνάντες. Θα μιλήσω και εγώ στα ισπανικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει ε, προκαταρτική ανάλυση των στοιχείων της αναφοράς αυτή και στη συνέχεια ήρθε και σε επαφή με τις αρμόδιες ισπανικές αρχές. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν δύο οδηγίες που πρέπει να εξεταστούν και να για τα ε, το πόσιμο ύδωρ και για τα λίματα, τα αστικά. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, όπως είχε πει και ο αναφέρον, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία που να ρυθμίζει την υδροδότηση. Ε, την παροχή ύδατος. Αυτό ε, έχει να κάνει ε, με τις προδιαγραφές. Δηλαδή η μόνη νομοθεσία που έχουμε ορίζει προδιαγραφές για την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχεται στους καταναλωτές. Ας πούμε το νερό πρέπει να είναι υγιεινό και καθαρή και να τηρεί κάποιες προδιαγραφές κάποιων μεγεθών και θα πρέπει το αρμόδιο κράτος να συμμορφώζεται. Σε μια προσφυγή επί παραλήψη, εξέτασε την οδηγία για τα λίματα στη συγκεκριμένη περιοχή και ε, σε σχέση με την απάντηση ε, των αρμοδίων αρχών μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής. Η πόλη αυτή λέει ε, ότι δεν έχει γίνει ειδικό ε, έλεγχος ειδική μελέτη για τις υποδομές και για τις αποχετεύσεις. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς πόλη, είναι ένας μικρός οικισμός εκεί η περιοχή ε, που είναι αποκομμένος μάλιστα και σε κάποια απόσταση από ένα αστικό κέντρο. Ε, μεσολαβούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, χωράφια κλπ. Οπότε, αυτό είναι μια αγρικία ας πούμε είναι 176 κάτοικοι σε αυτόν τον οικισμό ε, που είναι ε, κάτι ε, με το οποίο διαφωνεί ο αναφέρον που λέει ότι ο οικισμός έχει 500 κατοίκους και δεν είναι έτσι μια δευτερεύουσα οικιστική περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με την οδηγία για τα αστικά λίμματα, οποιαδήποτε πόλη ή οικισμός έχει κάτω από 2.000 κατοίκους δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ούτε καν χρειάζεται ας πούμε ένα σύστημα συλλογικής αποχέτευσης, υπόνομο δηλαδή, ο καθένας θα μπορούσε με ένα ιδιωτικό βόθρο ή κάποια συστήματα να φροντίζει την αποχέτευσή του. Καλό θα ήταν λοιπόν να αποταθεί στι αρμόδιε ισπανικέ αρχέ αναφέρων, που είναι περισσότερο αρμόδιε ακριβώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Γιατί ουσιαστικά είναι ελάχιστη, για να μην πω ανύπαρκτη, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής ε, Νομοθεσίας, κείμενης νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Δύο βουλευτέ έχουμε, να δούμε ποιο θέλει το λόγο. Really? είστε σίγουροι. Απίστευτο. Συνήθως έχω πάρα πολλούς βουλευτές που ζητούν το λόγο και έχουμε πρόβλημα χρόνου. Σήμερα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα κατά τη γνώμη μου. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν διαδικασίες επί παραβάση τρέχουσες κατά της ε, Ισπανίας από πέρσι, τον Οκτώβριο δεν απατώμε. Μήπως νέα αξιολόγηση, νέα μελέτη, έτσι πιστεύω. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Όπως σωστά είπατε, να απευθυνθούμε στις αρμόδιες περιφερειακές εμπροκειμένου αρχές και να στείλουμε επιστολή ε, και αυτή τη στιγμή ε, γίνει αυτό ως συνέχεια να κλείσουμε την αναφορά. Λοιπόν, θα στείλουμε ε, μια επιστολή με βάση τα όσα ακούσαμε σήμερα και τα λοιπά. Και μετά να κλείσει φορά. Γιατί εδώ πρόκειται για άλλο επίπεδο συνεννόηση με τις αρχές. Ωραία, τώρα γίναμε τέσσερις βουλευτές που παίρνουμε αυτή την απόφαση και συμφωνούμε όλοι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα ζήτημα χρόνου και περιμένουμε για την επόμενη αναφορά 606 ε, ε, σχετικά με τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση της παραβίασης οικονομικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. Ο κύριος Ροντρίγκες, κυρία Ροντρίγκες μάλλον είναι η αναφέρουσα, η οποία δεν έχει ακόμα καταφτάσει. Α, είναι στην είσοδο. Ε, επειδή τελειώσαμε νωρίτερα τα προηγούμενα, τι να κάνουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, 3-4-5 λεπτά, να κάνετε κανένα τηλεφώνημα και θα ξαναρχίσουμε. παρατέταρτο. Τέσσερις παρατέταρτο, όχι πέντε παρατέταρτο. Δεν κάνουμε μία ώρα διάλειμμα, κάνουμε ε, λίγα λεπτά. Πιείτε λίγο νεράκι, πείτε τίποτα με το γείτονά σας, αγοράστε καμιά μπανάνα, πάρτε καμιά βοηθό σας τηλέφωνο. Έχετε πέντε λεπτά όμως. Άντε και λίγο παραπάνω. Sharp in this room.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 Okay. I gave you a few minutes just... Ωραία, σας έδωσα μερικά λεπτά. Και τώρα προχωρούμε. Με χαρά καλωσορίζω την... τον Μαρτέρο Τρίγες, εκπρόσωπο της αναφέρουσας, καλωσορίσατε στην Επιτροπή Αναφορών ε, και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σας δίνω μέσα στο λόγο. Και παρακαλώ οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων να κάνουν ε, συζητήσεις εκτός της αισθούσης. Παρακαλώ, ησυχία κάνετε. Αν θέλετε να συνομιλήσετε έξω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροντρίγκε, έχετε το λόγο. Μπορείτε να μιλήσετε και γαλλικά και οποιαδήποτε άλλο από τι 22 επίσημέ μας ε, γλώσσε. Ε, η πρόεδρο το προτιμούσε σου ειδικά, αστείευαμε. Αλλά βεβαίω και αγγλικά και ισπανικά και γαλλικά. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Θα σας παρακαλέσω όμως να τηρήσετε το όριο το χρονικό των 5 λεπτών. σα έχουμε και το ρολόι για να σα βοηθάει. Σα ευχαριστώ. Είναι τιμή μου Βρίσκομαι στη συνεδρία σα εδώ σήμερα για να ακουστεί η φωνή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένειά μου αλλά μέσω αυτών και να, να ακουστεί και η φωνή του λαού από τη χώρα από την οποία προέρχομαι. Προέρχομαι από τον Μπενίν, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής. είμαι παντρεμένος, έχουμε παιδιά. Η, η γυναίκα μου είναι Γερμανίδα, γερμανική ηθαγένεια. Τα παιδιά μου έχουν δύο διπλή υπηκότητα, γερμανική και ελβετική και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Μπενίν. Σήμερα όμως βρισκόμαστε να έχουμε πέσει θύμα μιας πολιτικής κατάστασης, μια πολιτικής δίωξης θα μπορούσα να πω. Και θα σας το εκθέσω περιληπτικά, μιας και δεν έχω πάνω από πέντε λεπτά. Από την οικογένειά μου ε, και ε, αποσπάστηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στον Και δεν είμαστε οι μόνοι αυτής της που, που έχουμε πέσει θύμα αυτής της ε, κατάστασης, της αρπαγής, της περιουσίας μας. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε πριν να έρθει στην εξουσία η τρέχουσα, η τωρινή κυβέρνηση και οποτεδήποτε κάποιος ήταν είτε αντιφρονώνεται στην αντιπολίτευση, είτε απλώς εκπροσωπούσατε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό συμφέρον, θα έβρισκε ένα τρόπο, θα έβρισκαν ένα τρόπο να σας αρπάξουν την περιουσία. Χωρίς καμία δυνατότητα προσφογής στην δικαιοσύνη. Φανταστείτε ότι ο προσωπικός νομικός σύμβουλος, δικηγόρος του Προέδρου μας έγινε Υπουργός Δικαιοσύνης, συνεχίζει να είναι ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο μέλος και το τελευταίο που μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι αυτό το πρόσωπο έγινε και πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου της χώρας. Με λίγα λόγια δηλαδή όλες οι δικαιοδοτικές αποφάσεις είτε πρόκειται για πολιτικά ζητήματα, είτε πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα, είτε για οικονομικά θέματα ε, όλα αυτά θα βρίσκονται πλέον στα χέρια και θα εξαρτώνται από την καλή διάθεση του Προέδρου και του στενού κύκλου του. Η επιχείρησή μας. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Γιατί τη στιγμή η οικογένειά μου έχει χάσει όλη της την περιουσία στο Μπενίν. Ε, ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, ξεροδοχειακές βάμβακος στην ε, Αφρική. Πέρυσι η οικογένειά μου έχασε 35, πάνω, πάνω περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ από συμβάσεις με τις οποίες είχαμε, τις οποίες είχαμε υπογράψει με την, ε, τον όμιλο Λουίντ Τρεφούς και τις οποίες δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε. Στο τρέχον οικονομικό έτος έχουμε χάσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν θα μπορούσα τώρα μέσα σε 5 λεπτά να σας εκθέσω όλες αυτές τις εξελίξεις, όλα αυτά τα γεγονότα. Αλλά ένα θα σας πω, Δημόσια δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας ότι για να επανεκλεγεί κανείς δεν χρειάζεται ένας καλός απολογισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί να καταπνίγει την αντιπολίτευση, να ε, καταπολεμά, να εξαλείφει αυτούς που τον ε, που του αντιτάσσονται. Και αυτό προσπαθεί να κάνει υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, φυλακιστεί. Ακόμα και βουλευτές έχουν μπει στη φυλακή. Ακόμα και οι αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου που είχαν ληφθεί πριν να έρθει στην εξουσία ο, τρε... ο σημερινός πρόεδρος δεν εφαρμόζονται. Ε, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου σας γιατί φτάσαμε στα πέντε λεπτά. Όμως τι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση γιατί η περιουσία μας είναι μεγάλη. Η περιουσία της, την οποία μας άρπαξαν είναι τεράστια. Πρόκειται για επενδύσεις πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα η οποία υποφέρει. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σακό ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ. Περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ γαλλικά. Διπλό το περιεχόμενο του αιτήματο που περιέχεται σε αυτή την αφορά. Από τη μία πλευρά ο αναφέρον θέλει μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διένεξη αυτή μεταξύ της, της οικογένειάς του και της κυβέρνησης του Μπενίν, της νέας κυβέρνησης με τον νέο πρόεδρο. Από την άλλη πλευρά όμως μας ζητήθηκε να καταφέρουμε να παρεύουμε κι εμείς στην κυβέρνηση αυτή προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο στη χώρα αυτή αλλά και σε υπόλοιπες αφρικανικές χώρες την ε, οικονομική και προσωπική περιουσία των ε, πολιτών υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εξετάσουμε με βάση πληροφορίες αυτές την αναφορά και να δούμε έπειτα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τη διένεξη της οικογένειας το αναφέροντος με την κυβέρνηση του Μπενίνης, η στασή ήταν η ακόλουθη το καλύτερο να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Μπενίν. Από όσο κατάλαβα από τις εξηγήσει σας, δεν εμπιστεύεστε ιδιαίτερα το δικαστικό σύστημα του Μπενίν. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να προσφύγετε στα περιφερειακά δικαστικά όργανα, όπως για παράδειγμα το Δικαστήριο της Δικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ή θα μπορούσατε να Απευθυνθείτε επίσης και στον Οργανισμό για την Αρμόνιση του Δικαίου των Επιχειρήσεων στην Αφρική. Αν το κάνετε αυτό, βέβαια η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον Πενίν θα είναι στη διαθεσή σα προκειμένου να καταφέρει να σα συνδράμει, προκειμένου να γίνουν αυτέ οι προσφυγέ σε αυτούς του περιφερειακούς οργανισμούς. Όσον αφορά όμω τώρα το δεύτερο σκέλος της αναφορά σα, δηλαδή την προστασία των δικαιωμάτων επενδυτών στην Αφρική, Ω προ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την νομική δικαιοσύνη, καθώς επίσης και στρέφεται κατά της ατιμορρησίας, προκειμένου να προωθήσει την επιχειρηματικότητα παντού. Και αυτό γίνεται με τρεις τρόπους. Έχουμε καταρχάς τον πολιτικό διάλογο που γίνεται με τις κυβερνήσεις εταίρους ε, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού, άρθρο 8 συγκεκριμένα. Από την άλλη έχουμε τον λεγόμενο περιφερειακό τομεακό διάλογο που γίνεται σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει και μια συνιστόσα βελτίωση επιχειρηματικότητας και τρίτον Έχουμε και το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 και ένας βασικός πυλώνας του εξωτερικού αυτοπενδυτικού σχεδίου είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που εξηγήσατε πώς έχει η κατάσταση. Ενδεχομένως να μπορούσαμε να ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους. Έχετε το λόγο. Κύριος Γιάρ. Τώρα μόλις ε, και κοιταζόμαστε με κάποια απόγνωση με τους συναδελφούς και απελπισία. Καταλαβαίνω την κατάσταση, ακούσαμε τι συμβαίνει και το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς πραγματικά να βοηθήσουμε. Είναι πολλά τα τεινά εδώ. Μιλάμε για την οικονομική ανάπτυξη, για το προσφυγικό, και όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι προσκρούμε στις πολιτικές καταστάσεις και σχετισμούς. δημοκρατία λαμβάνει πολλές ε, μορφές, αλλά δεν σημαίνει πάντα και κράτος δικαίου. Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία γενικότερα, η οποία δεν είναι δεδομένη εδώ. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τον αναφέροντα. De facto δηλαδή το έχουν δημεύσει την περιουσία στη χώρα αυτή επειδή άλλαξε ο πρόεδρος, ε, μας λέει ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να επιβάλλει το κράτος δικαίου. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει, ε, να σου συμβεί τέτοιο πράγμα. Και γι' αυτό κοιτάω και τους συναδέλφους πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Έκανε κάποιες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το πιο αποτελεσματικό ποιο θα ήταν. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εμεί οικονομικές σχέσεις με τον Μπενίν και μπορούμε να πιέσουμε. Η πρώτη πρόταση ήταν μια διαδικασία διαβούλευσης με τη χώρα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχουμε οικονομικές σχέσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά. Και μετά είναι το κράτος δικαίου. Κάτι που με ενοχλεί και, και με έχει εκνευρίσει τώρα γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε. Και εγώ είμαι γεωργός και ξέρω τι σημαίνει ιδιοκτησία. Και ξέρω ότι σήμερα ακόμα περισσότερο γιατί έχω μεγαλώσει τον κομμουνισμό, ότι σημαίνει να σου παίρνουν την περιουσία και να μην έχει και καμία προσφυγή, κανένα καταφύγιο πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Anybody else? Θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε νομίζω καλά την κατάσταση. Ε, κύριε Ροντρίγκε, ε, η υπόθεσή σας, η κατάστασή σας μας ε, συγκινεί όλους. Έχετε συνεισφέρει πάρα πολύ στην περιοχή, έχετε δώσει εργασία σε πάνω από χίλιους ανθρώπους, ανθρώπους που υποφέρουν, που έχουν να αντιμετωπίσουν την ανεργία και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το λοιμό. Επομένω, η συνεισφορά σας είναι πολύ σημαντική και την αναγνωρίζει η Επιτροπή μας. Θεωρούμε πολύτιμη και σας ευχαριστούμε για τι τις προσπάθειες, τις ε, θαραλέες που κάνετε. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο πάλι για να απαντήσετε σε αυτά που ακούσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτά που είπε ο συνάδελφος. Και να σας πω ότι υπάρχει το χρονικό όριο, αλλά μην ε, προσπαθείτε τόσο πολύ να περιοριστείτε όπως πριν. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έβλεπα τηλεόραση και άκουσα τη συνέντευξη τύπου της ε, καγκελαρίου Μέρκελ που μιλούσε για τα θέματα του μεταναστευτικού στην Αφρική. Και για μια άλλη φορά θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να σας ομιλώ σήμερα. Υπάρχει κάτι που με ταλανίζει και με βασανίζει. Και είναι απλό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η Αφρικανική Ήπειρος που υποτίθεται ότι είναι η πλουσιότερη από πλευράς φυσικών πόρων να παράγει μόνο μετανάστες και πρόσφυγες από τη βία και τον πόλεμο. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν δώσετε μια μικρή επικράτεια σε έναν Αφρικανό, την χρησιμοποιεί για να καταστρέψει τους συμπατριώτες του σήμερα έχουμε μια κατάσταση που είναι απέναντι στις ίδιες τις αρχές και τις αξίες σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, καταπολεμάει τα μονοπόλια, για να μην αναφέρω τίποτα παραπάνω οικονομικά. Σήμερα στον Πενίν, όμως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ελέγχει 100% το κοινοβούλιο. Στι 2 η ώρα το πρωί με 10-12 βουλευτέ μπορούν να περάσουν ένα νόμο που θα αλλάξει τα πάντα στη χώρα. Και υπάρχουν και αποδείξεις γι' αυτό. Είναι πρόεδρο τη λιμενική αρχή, ελέγχει με τι εταιρείε του το λιμάνι, το, τα, τον αερολιμένα, το βάμβακα, τα λοιπάσματα, ε, ε, τη γεωργία, τη δικαιοσύνη, όλα τα ελέγχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στέλνει ε, σημαντική βοήθεια για την καταπολέμηση αυτής της φτώχειας που οδηγεί στη μετανάστευση. Και τους ανθρώπους αυτούς που ξεβράζει η θάλασσα στις ακτές σας και πεθαίνουν εδώ. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Εγώ δεν έχω τίποτα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μου λέει να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μας φάγανε όλα τα λεφτά οι δικηγόροι. Δεν έχουμε τώρα χρήματα για να πληρώσουμε δικηγόρου. Έχουμε στερέψει και δεν έχουμε και ενέργεια για να παλέψουμε. Επίδε το κάνουνε, εσκεμένα, ε, σε στραγγαλίζουν, σε γονατίζουν. Ο δικαστής που αποφάσισε να μας αρπάξει το εργοστάσιό μας που αξίζει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ. Αρνήθηκαν να αποτιμήσουν, να κάνουν μια εκτίμηση για την αξία. Τελείω αυθαίρετα το ε, κατάσχεσαν. Και εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε αναμοχλοποίηση, συνεργάζεστε με τις χώρες και τις αφρικανικές χώρες, ακριβώς στο πλαίσιο των χωρών ε, Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού. Έχετε πολλά προγράμματα, έχετε και αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τόπου. Κάθε μέρα συνεργάζεστε σε επιτροπές για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι πολύ μοχλή και τα μέσα πίεσης ο πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού ζήτησε να μεσολαβήσει ανάμεσα στη δική μας επιχείρηση και την κυβέρνηση του Μπενίν. Ατελέσφορο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας Αφρικανός ηγέτης να πάει να δει έναν άλλον Αφρικανό ηγέτη και να του πει ε, μη βασανίζεις την αντιπολίτευση. Γιατί δεν θέλει να πάει να του πει το ίδιο για τη δική του χώρα κάποιο άλλο ηγέτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν που είναι εκτός Αφρικής μπορεί να δράσει. Αν εμεί κάναμε κάτι λάθος, να μα το πείτε αν η οικογένειά μου έχει σφάλει κάπου. Εμείς ζητάμε τη βοήθειά σας και σε νομικό επίπεδο. Κοιτάξτε, παληθεύστε αν ευσταθούν αυτά που λέμε ή αν ισχυριζόμαστε διάφορα ψεύδι. Ελέγξτε το. Και πραγματικά γονατίζουμε μπροστά σας και σας, σας εκλυπαρούμε να εμπλακείτε. Και μέχρι τέλους. Είναι πολιτικό το πρόβλημα. Και δεν είμαστε μόνη περίπτωση εμείς στον Πενίν. Πώς είναι δυνατόν να ανταγωνιστείς την εταιρεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και να κερδίσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε να πάω να δω ποιον δικαστή θέλετε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά δεν θέλω να σας ε, καταχρωστώ όλο το χρόνο. Αλλά σας παρακαλώ, κοιτάξτε το, ε, ερευνήστε το μέχρι τέλους. Για να δείτε και η ίδια η δράση που κάνετε εσείς, κατά πόσο σαμποτάρετε και υπονομεύετε από τέτοιες συμπεριφορές. Έχετε ε, κατατάξει ως δημοκρατική χώρα τον Μπενίν. Για πηγαίνετε εκεί παρακαλώ να δείτε τι γίνεται. Είναι δραματική η κατάσταση. Οι συνδικαλιστές, οι πάντες έχουν γονατίσει, τους έχουν γονατίσει. Τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Κανείς δεν έχει κανένα δικαίωμα πλέον στον Μπενίν. Και δεν έρχομαι αυτά να σας τα πω εδώ βάλτε το όνομά μου στο, στο Google να δείτε πόσες φορές έχω καταγγείλει ε, τη διαφθορά. Είμαι επιχειρηματίας, δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες διαφθαρμένοι. Μπορεί κανείς ε, με έντιμο τρόπο και ειλικρινή και τα, τη, ζωή του να κερδίσει και να πλουτίσει. Και η οικογένειά μου δεν έκανε τίποτα για να αξίζει τέτοια συμπεριφορά. Τα παιδιά μου, η σύζυγός μου, γιατί δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Μα προφανώς δεν κάνετε τίποτα για να αξίζετε μια τέτοια μοίρα. Ωστόσο όμως η δική μας η Επιτροπή μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, σίγουρα ναι, αλλά ας ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί τρόπον την η κατάσταση, ότι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής όμως, οι μέθοδοι και οι δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και θα προσπαθήσω τώρα να συνοψίσω και την όλη συζήτηση και ελπίζω ότι έχω την υποστήριξη των συναδέλφων αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχάς σας ενθαρρύνουμε να απευθυνθείτε στον Οργανισμό για την Εναρμόνιση του Δικαίου των Επιχειρήσεων στην Αφρική και στο δικαστήριο και διαιτητικό δικαστήριο προβλέπει αυτός ο οργανισμός. Νομίζω ότι από τη διαιτησία θα πρέπει να περάσετε. Σας ενθαρρύνουμε πραγματικά να περάσετε από τα περιφερειακά αυτά δικαστικά όργανα, τα οποία μπορεί πραγματικά να ασχοληθούν με την επίλυση της διαφοράς αυτής μέσω της διαιτησίας και ενδεχομένως να οδηγηθείτε έτσι και σε αποζημίωση για όλα αυτά τα οποία έχετε υποστεί. Θα έλεγαν συνεχεία ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε ως Επιτροπή μία επιστολή ενημερωτική στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Μογκερίνη δηλαδή, προσπαθώντας εκεί να της εξηγήσουμε πώς έχει η κατάσταση και ποιες είναι οι ανησυχίες που έχουμε όσον αφορά την κατάστασή σας στον Μπενίν, κύριε Ροντρίγκε. Γιατί πραγματικά η κατάστασή σας είναι δεινή, πολύ σοβαρή και όντω αναφέρεστε εδώ πέρα σε γεγονότα, φαινόμενα τα οποία είναι συστηματικά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με εσά, με τη δική σας προσωπική κατάσταση. Λοιπόν, Α κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ πάντω ότι ω Επιτροπή Αναφορών δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε δικαιοδοσία στον Πενίν. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να τονίσει και να υπογραμμίσει μόνο την κατάσταση με διαφορετικών μέσων, αλλά εκεί περιορίζεται η αρμοδιότητά μα. Εν συνεχεία, θεωρώ ότι θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή, γιατί θα έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να κάνουμε και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω και βλέπω ότι γνέφουν θετικά οι συνάδελφοι. Ο Πίτερ Γιάρ, παρακαλώ. Έχω μια σύντομη συμπλήρωση μόνο. Γιατί γνωρίζω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού γίνονται πάρα πολλέ συζητήσεις ακριβώς για αυτό το θέμα, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Να δούμε τι την κάνουν όμως για την αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχει διαφθορά και, κάτι, και ένας δεύτερος παράγορα, έτσι, πολιτική πίεση. Και δεν γίνονται και έλεγχοι για τα ασφάλματα της εκτέλεσης ε, αυτών των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Πραγματικά τονίζω ότι θα πρέπει να γίνει διάλογος. Αν δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια στον Πενή, να θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να κάνουμε και ένα πολιτικό διάλογο, όχι μόνο οικονομικό. Δηλαδή να στέλνουμε λεφτά και εντάξει και ελπίζω να πιάνουν τόπο. Εντάξει, τα λέω λίγο χοντρά και υπερβάλλω. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε το διάλογο αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κατά τα άλλα, έχει απολύτω δίκιο η πρόεδρο. So, actually. Μάλιστα, λοιπόν, θα κινηθούμε όπω περιέγραψα. Τρία διαφορετικά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Ήδη σα εξήγησα αυτά τα οποία είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς μπορούμε να κινηθούμε όσον αφορά το κοινό και διαιτητικό δικαστήριο του Οργανισμού για την Αρμόνιση του Δικαίου των Επιχειρήσεων στην Αφρική, πρώτον αυτό, και δεύτερον θα αποστείλουμε μία επιστολή στην ύπατη εκπρόσωπο, θα προωθήσουμε επίση την αναφορά αυτή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και εν συνεχεία πραγματικά θα έχουμε εξαντλήσει εντελώ τα δικά μα τα μέσα τι δικέ μα δυνατότητε και θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Για άλλη μια φορά, πάντω, ε, σα ευχαριστούμε, κύριε Ροντρίγκε, που ήρθατε εδώ για να μα μιλήσετε για εσά τον ίδιο, για την οικογένειά σα, για την επιχείρησή σα και εν γέννη για όλου αυτού του ανθρώπου που πλήττονται από την πολύ αυτή δύσκολη κατάσταση. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά τα οποία σα περιέγραψα και ελπίζω ότι μακροπρόθεσμα θα αποβούν θετικά για σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σε Βρυξέλλε σήμερα και όπω σα είπα, θα κάνουμε κάθε το δυνατό για να σα βοηθήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Θα κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε καταφέρει να κινηθούμε πιο γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Πάντως, μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της. Δεν είναι οι αναφέροντες, είναι ήδη παρόντες στην αίθουσα. Αναφέρομαι στην αναφορά 0607 σχετικά με τις μειώσεις των ισχύσεων για τη βιολογική γεωργία. Οι αναφέροντες είναι εδώ, μαζί μας και έχουν και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση PowerPoint, έτσι δεν είναι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Άντρες Γκαρθία Βακέρο, καθώς επίσης και τον κύριο Φελίπε Αβίλα Γκονζάλες. Έχετε το λόγο για μερικά λεπτά, για 5-6 λεπτά. Καλησπέρα σας. Άντρες Γκαρθία λέγομαι ε, και ο Φελίπε Άβελα μαζί μου από τις οργανώσεις πολιτών στη Καστία Λαμάτσα στην Καστήλη ε, Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μα δίνετε. Η οικολογική γεωργία, βιολογική γεωργία δεν είναι βιώσιμη οικονομικά. Γι' αυτό υπάρχουν κρατικέ ενισχύσει στο πρόγραμμα ανάπτυξη τη υπαίθρου. Το πρόγραμμα αυτό είναι υπό την επίβλεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητά βοήθεια υπογράφοντα μία σύμβαση. βοήθεια δεσμευμόμαστε ότι επειδή μία σύμβαση όπου οι αγροτε δεσμευόμαστε ότι επί μία πενταετία θα έχουμε βιολογική γεωργία. Αυτή η ενίσχυση ζητήθηκε το Μάρτιο του 2015 από την Καστήλη Λαμάντσα και αργότερα το 2016 όταν είχαμε σπείρει ήδη δύο χρόνια από τα πέντε η τοπική κυβέρνηση της Καστήλης Λαμάντσα αναδρομικά άλλαξε ε, τα ποσά και μείωσε κατά 67% τις ενισχύσεις. Ε, αυτό είναι ε, αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού στα μέσα του παιχνιδιού. Άρα 3.297 γεωργοί, που είναι περίπου η μισή βιολογική γεωργοί, ε, πετάχτηκαν έξω από αυτό το σχήμα. Την περασμένη Παρασκευή σας στείλαμε όλα τα έγγραφα της περιφερικής κυβέρνησης σχετικά με την ενίσχυση και θα δείτε ότι τίθεται θέμα εύλογη εμπιστοσύνη και ασφάλεια δικαίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα σχετικά. Ε, Σα έχουμε ένα πίνακα εδώ με ε, χρονολογική σειρά. Αναφέρονται τα διάφορα έγγραφα, τα βλέπετε εδώ, ε, που έχουν ε, εκπονηθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Περιφερειακή Κυβέρνηση. Η Περιφέρεια τη Καστήλη Λαμάντσα ζήτησε στι 25 Ιουλίου 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει το πρόγραμμα βιολογικής ε, γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έτυχε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ήταν σωστό θα είχε εγκριθεί ως είχε. Αλλά δεν είναι 100% σωστό, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να αναθεωρηθεί και να είναι το άθροισμα τη αρχική πρόταση συν τη τροποποίηση, Πράγμα που δεν έγινε. Και θα πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν συνέβη αυτό. Και τελικά το σχέδιο ανάπτυξη τη υπαίθρου που εγκρίθηκε επιτράπει να γίνουν τροποποιήσει που δεν είχαν συμπεριληφθεί στι παρατηρήσει. Το Νοέμβριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί τι παρατηρήσει τη στην πρόταση και δεν είναι απλώ ένα προσχέδιο αυτό. Δεν υπάρχει καμία ε, πρόταση που να λέει ότι τα ποσά δεν είναι τα σωστά. Και στον επόμενο πίνακα θα δείτε τις ενισχύσεις και τα ποσά και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και της Περιφερειακής Κυβέρνησης. Τι διαπιστώνουμε από τον Ιούλιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε τα ποσά να μειώνονται 20% τον Αύγουστο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2015 67% στο τελικό κείμενο που εγκρίθηκε για την ανάπτυξη Πέθρου. Αργότερα η τοπική κυβέρνηση λέει ότι συνάδει με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία η πρότασή της και με τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε δεν χρειάζεται εκ των υστέρων καμία τροποποίηση. Επίσης λέγουν ότι η ενίσχυση ε, έχει και ανασταλτικό όρο μέχρι να εγκριθεί το πρόγραμμα, δηλαδή δεν θα μπορούσαν ούτε να εγκριθούν ούτε να εκταμιευθούν οι ενισχύσεις. Ε, υπήρχε και μια άλλη διάταξη για, με ανασταλτικό χαρακτήρα που δεν εγκρίθηκε τελικά γιατί ήταν ε, παράνομη. Επίσης, ο, προ, ο υπολογισμός σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής επιτρέπεται και εγκρίθηκε να αυξηθεί κατά 17% ε, χωρίς να μειωθούν ε, τα ποσά τον ε, Ιανουάριο του 2016 η τοπική κυβέρνηση όταν είχε λάβει όλες τις αιτήσει γιατί είχε εκνέψει η προθεσμία ε, εδώ και 9 μήνες και πλέον, βγάζει μια έκθεση με τέσσερις υποθέσεις για επαναυπολογισμό των ποσών. Και με τρόπο αυθαίρετο άλλαξε τα ποσά, της ενισχύσεις, χωρίς καμία τεκμηρίωση και δικαιολογία και ε, διαταράσει και διαρριγνεί και την ασφάλεια δικαίου και τις σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής πίστης. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό τώρα. Δεν μπορεί, ε, όταν δίνεις εξετάσεις κρατικές για να πάρεις ένα πτυχίο, δεν μπορούν να αλλάζουν στη μέση των εξετάσεων τους όρους και τις προϋποθέσεις. Υπάρχει και απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ε, που ορίζει ότι δεν μπορούν να μειώνονται έτσι αυθαίρετα τα ποσά, αλλά στη συνέχεια δικαιολογεί τη μείωση, διότι λέει ε, εκτελείται απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η μείωση των ενισχύσεων οδήγησε ε, στο να είναι αφόρητη και αβίωτη και μη βιώσιμη δηλαδή η βιολογική γεωργία, ούτε οι εκτάσεις που έχουν προβλεφθεί. Η περιφερειακή κυβέρνηση δίνει 400 εκατομμύρια για τα δάση. Από την εταιρεία Χιακάν, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ε, εκταμίευση ενίσχυση σε περιφέρεια. 6, 7, 8 λοιπά ε, ε, του κανονισμού 1303 ε, του 2011 έχουν γίνει σεβαστά και η αρχή της ασφάλειας δικαίου και τα λοιπά επίσης γίνονται σεβαστά. Ζητούμε να γίνει έλεγχος ε, λογιστικός σε αυτά τα 400 εκατομμύρια που έχουν δώσει για τα δάση και να αλλάξει η κατάσταση και να μπορέσει να διατηρηθεί στην Καστήλη Λαμάντσα η βιολογική γεωργία υπέρ ε, της δημόσιας ε, υγείας και υπέρ του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. This... Και εμείς σας ευχαριστούμε. Η αναφορά σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Παρευρίσκεται επίσης εκπρόσωπος της περιφέρειας της Καστήλης Λαμάντσα Πιλάρ Ζηλανδράδο, η που κάθεται εκεί και θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Μάλιστα, τώρα λειτουργεί το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση της Καστήλης Λαμάντσα και θα ήθελα να προσθέσω μερικά στοιχεία προφορικά πέρα από τα γραπτά που σας έχουμε στείλει για την βιολογική γεωργία και να καταλάβουμε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και την αναφορά. Τι γίνεται στην περιφέρειά μας. Πρόκειται για εξορθολογισμό και για μεγαλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ε, ευθύνη. Το Μάρτιο του 2015 εγκρίθηκαν κάποιες ενισχύσεις, αλλά αυτές συνδέονταν και ήταν υπό την αίρεση της έγκρισης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Αυτό μέχρι τότε δεν είχε ολοκληρωθεί, άρα έπρεπε να κλείσει ε, ο προϋπολογισμός ε, με διάφορα μέτρα ε, εξισορροπημένα στους διάφορους κλάδους γιατί υπάρχουν και κοινοτικές προτεραιότητες. Στην προηγούμενη περίοδο 2007-2013 είχαν εγκριθεί 6.510 αιτήσει βιολογικής γεωργίας και από τα 38.000 εκτάρια είχαν επταπλασιαστεί οι ε, γέες το 2014 και μια απλή ε, αριθμητική πράξη καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε όλες αυτές τις αιτήσει με τις ίδιες ενισχύσεις αφού είχαν επταπλασιαστεί. Βασικός στόχος των ενισχύσεων είναι η διατήρηση και η βελτίωση των γεωργικών οικοσυστημάτων. Στόχος λοιπόν είναι να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια στη βιολογική ε, παραγωγή. Οπότε, επειδή οι κλιματικές ε, και οι κλιματολογικές συνθήκες στην Καστήλη ε, Λαμάντσα ευνοούν τη βιολογική ε, καλλιέργεια ε, για το αμπέλι, για την ελιά και για κάποιες άλλες καλλιέργειες οποροκυπευτικών ε, έχουν εγκριθεί κάποιες ενισχύσεις σε σχέση με τις πραγματικές τιμές για να αντισταθμιστεί η απώλεια εισοδήματος. Και είναι και περισσότερη η παραγωγή και περισσότερα τα εκτάρια. Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης ε, και έχουν υποβληθεί αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 214 εκατομμύρια ευρώ, 14% της συνολικής δημόσιας δαπάνης προβλέπονται για ένα και μόνο μέτρο του προγράμματος. Και η πρώτη τροποποίηση έγινε τον Απρίλιο του 2017, όπου προσθέθηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από άλλες γραμμές του προπολογισμού που μειώθηκαν και τελικά η βιολογική γεωργία πήρε 253 εκατομμύρια ευρώ σύνολο, ίσον 16% των δημοσίων δαπανών της περιφέρειας, που σημαίνει αύξηση περίπου 20% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Σε σχέση λοιπόν με όλα αυτά, ε, δημοσιεύτηκαν και άλλα έγγραφα το 2016 και το 2017. Εγκρίθηκε ε, ε, μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων 8.089 και η βιολογική γεωργία καλύπτει 326.000 εκτάρια. Στην Καστήλα Μάντσα. η βιολογική γεωργία είναι προτεραιότητα για τον αγροδιοτροφικό τομέα της περιφέρειας και για την κατανάλωση τέτοιων προϊόντων. Οπότε μπορεί κανείς να συναγάγει ότι παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες και περιορισμούς που έχουμε από την κρίση, στηρίζουμε τη βιολογική γεωργία, είναι προτεραιότητά μας στην Καστήλη Λαμάντσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The commission is still... Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσωπείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πάντα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Έμπρετς Θα μιλήσω γαλλικά. Να αξιοποιήσω και τους διερμηνείς. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε ε, ήδη συζητήσει για το θέμα, είχαμε ήδη συναντηθεί και δεν ε, διαπιστώνω να υπάρχει κανένα νέο στοιχείο. Ε, διαπιστώσαμε και τότε ότι είχαμε διαφορετικές θέσεις και αντιλήψεις της κατάστασης. Ε, το διαπιστώνουμε και σήμερα. Εγώ θα παρουσιάσω την αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης Καστήλης Λαμάντσα εγκρίθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2015 και κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οτιδήποτε είχε συμβεί πριν από εκείνη την ημερομηνία δεν δεσμεύει ουδόλως την Επιτροπή. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ζωντανό και έχει υποστεί διάφορες τροποποιήσεις όπως πάντοτε συμβαίνει με τα προγράμματα αυτά. Ε, ωστόσο η κατάσταση είναι εξαιρετικά απλή. Λάβαμε ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το 2014 και το οποίο ήταν χαοτικό. Δεν μπορούσαμε να το θεωρήσουμε αξιόπιστο. Γι' αυτό το λόγο στείλαμε ε, στην περιφέρεια μια επιστολή η οποία πράγματι στις 13 ε, Νοεμβρίου του 14 απεστάλλει. Επί τη βάση λοιπόν αυτής της επιστολής, η οποία είχε 329 ε, παρατηρήσεις, το Ρίστον παραδό και αυτό σας δίνει μία αίσθηση της ποιότητας του σχέδιου που είχαμε λάβει, θα, καθίσω, θα, σταθώ στο 242, στην παρατήρηση 242 με την οποία διαψεύδουμε μία από τις, α, από τις, τους ισχυρισμούς των αναφερόντων που λένε ότι δεν είχαμε αναφέρει τίποτα σε σχέση με τα ποσά. Δεν είχαμε πράγματι ε, διαφωνήσει με το ποσό. Γιατί δεν είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σχολιάσει το συγκεκριμένο ποσό. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να σχολιάσει τη μεθοδολογία με την οποία η περιφέρεια καταλήγει σε αυτό. Και θα συνεχίσω στα ισπανικά. Λέγαμε λοιπόν ότι ε, θα ε, ισχύουν ε, οι διατάξει του άρθρου 10 του κανονισμού 808-2014 με βάση αναφοράς του υπολογισμού των των ενισχύσεων. Πάντα μιλάω στο μέλλοντα όμως και θα βασιστεί σε μία μέθοδο αξιολόγηση των απολειών εισοδήματος και του επιπλέον κόστος που απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης. Και η, τιμή καταναλωτού ε, που θα είναι ελαφρώς αυξημένη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό και αυτό θα βασιστεί στα πιο πρόσφατα στοιχεία ε, από ένα όργανο αρμόδιο ε, με πιστοποίηση. Όταν τα λέμε όλα αυτά, τι σημαίνουν. Ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το παραμικρό ποσό ενίσχυση στη βιολογική γεωργία, τα περιβαλλοντικά μέτρα ή οτιδήποτε άλλο μέτρο αντισταθμιστικό, σε περίπτωση που δεν βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία τεκμηριωμένη και κοστολογημένη και το πρόγραμμα όντως που μας υπέβαλαν κατά το θέρος του 2014 δεν έλεγε τους τίποτα σχετικά. Οτιδήποτε. Ήταν απλώς στοιχειώδες που δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε ε, ως ε, μη σοβαρό. Δεν σχολιάσαμε λοιπόν κάτι το οποίο δεν άξιζε να σχολιαστεί. Μετά, η αρχή διαχείρισης δημοσιοποίησε, έκανε προκήρυξη οι αιτήσει. Όμως αυτό έγινε πριν από την έγκριση της, ε, του προγράμματο, δηλαδή την 30 Οκτωβρίου 2015, επομένω δεν τον γνωρίζουμε και δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω μπορεί αυτό να οδηγήσει σε διαμαρτυρίε στην Καστήλη Λαμάντσα και γνωρίζουμε ότι για αυτούς τους λόγους η περιφερειακή κυβέρνηση χρειάστηκε να αναθεωρήσει ορισμένες από τις λεπτομέρειες και ιδιαίτερα όσον αφορούσε τις ε, βιολογικές καλλιέργειες έγιναν τροποποίησεις. Οι τροποποίησεις αυτές δεν ικανοποιούν τους ετούντες, οι οποίοι θα ήθελαν έναν ουσιαστικά μεγαλύτερο κονδύλι, έναν ουσιαστικά αυξημένο προϋπολογισμό για τη βιολογική καλλιέργεια και να φτάναμε ουσιαστικά στο ποσό το οποίο προέκυπτε από την ε, προκήρυξη του 2015. Ε, σας εξέθεσα πώς και σας το, επαναλάβω, εκτιμά ότι έχει κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ο ρόλο τη να ε, εκφράζει κάποια άποψη σε σχέση με το ύψο των ποσών. Εκφράζουμε ε, άποψη σε σχέση με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν τα ποσά αυτά. Κάτι ακόμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε και είναι προς ε, υπέρ της θέσεως μάλλον της Καστήλης Λαμάντσα είναι ότι το μέτρο αυτό κινητοποιεί το 14% των συνολικών δαπανών του προγράμματος τους, ενώ στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6%. Επομένως δεν μπορεί κανείς να δεχθεί τον ισχυρισμό και την κατηγορία ότι η Καστήλη Λαμάντσα δεν υποστηρίζει τη βιολογική καλλιέργεια. Τώρα, τον Απρίλιο του 2017 λάβαμε ε, επί τη βάση μιας πρότασης του, από το φθινόπωρο του 2010, ε, την πρόταση να προσθεθούν και άλλα 20 εκατομμύρια πέραν εκείνων που είχαν προβλεφθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, φτάνοντα ένα σύνολο 235 εκατομμυρίων ευρώ. Και ε, το στοιχείο στο οποίο σταθήκαμε δεν είναι τόσο το ύψος του ποσού, αλλά το ότι θα πρέπει να αναλυφθούν δεσμεύσεις επί τη βάση των αποτελεσμάτων που θα έχει το πρόγραμμα. Δηλαδή, οι αρχές της Καστήλης Ναμάντσα θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αυξηθεί η ε, ε, έκταση η οποία ε, επηρεάζεται από αυτά τα μέτρα, δηλαδή να πάει στα 366.000 εκτάρια από 258.000 που ήταν στην αρχική πρόταση και αυτό ήταν το πολιτικό στοιχείο στο οποίο επιμείναμε. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο καλοκαίρι, ότι θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι προγράμματα τα οποία προσπαθούν να ε, ε, βοηθήσουν τους αγρότες. Είναι προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν το περιβάλλον και είναι κάτι στο οποίο επιμένουμε. Και συγχωρήστε μου την έκφραση, αυτά τα μέτρα δεν είναι σεξι. Υπό την έννοια ότι δεν είναι σχεδιασμένα για να ε, προσφέρουν συμπληρωματικό εισόδημα στους αγρότες που έχουν απώλειες. Είναι, ε, υπάρχουν δυνατότητες ε, τέτοιες σε άλλα μέτρα, όμως μιλούμε για μια περιφέρεια η οποία έχει σημαντικές απώλειες, ίσως μεταξύ άλλων της παραγωγικότητας της συνολικής που, που επιδεικνύει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μπορούν οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Υπάρχει ένα κατάλογο ομιλητών. Η κυρία Γιούσον η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τους αναφέροντες στην κυβέρνηση της Καστήλινα Μάντσα και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Η αγρότες στην Καστελίνα Μάντσα αντιμετωπίζουν ε, μια κατάσταση που δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Έχουν δεσμευθεί επί πέντε χρόνια να καλλιεργούν με βάση κάποιες προϋποθέσεις και όταν άρχισαν λοιπόν να σπέρνουν και να καλλιεργούν ε, μειώθηκαν οι ενισχύσει κατά 67%. Μιλούν για έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Η κυβέρνηση τη περιφέρεια Καστήλη, Λαμάντσα μα μιλά για ποσότητε και για επιφάνειες, ε, για στρέμματα και εκτάρια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας μιλάει για τα κριτήρια που είναι τα εφαρμοστέα και που εφαρμόζονται. Αλλά όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να διαρευνούμε για ποιο λόγο άλλαξαν αυτά. Μπορεί να είναι καλή ή κακή η διατύπωση και η ρύθμιση του σχεδίου του αναπτυξιακού που έχουν υποβάλει. Ε, αλλά χωρίς να γίνουν ε, κάποιες προτάσεις ή αμφισβητήσεις ε, και προτάσεις για βελτίωση, το μειώνουν κατά 67%. Πραγματικά είναι πρόβλημα ανασφάλειας για τους καλλιεργητές τους ε, βιολογικούς. Και θέλω επίσης επ' ευκαιρία να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην έχουμε ε, προβλήματα να έχουμε ε, κατευθυντήριες γραμμές για να μην συγκρούονται μεταξύ τους οι ε, αυτόνομες περιφέρειες. Γιατί στη, ε, στην Ισπανία αυτές είναι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στις περιφέρειες. Και αν δεν έχουμε γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ, υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Γιατί δεν είναι το ίδιο να είσαι καλλιεργητή βιολογικό σε μια ή άλλη περιφέρεια. Γιατί τέτοια δραστική αλλαγή, περικοπή 67%, 67% είναι πολλά τα λεφτά για να μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει έτσι με μια μονοκονδυλιά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. Gutierrez. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκουτιέρες πρέπει έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο προφανώς είναι από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου υπάρχει αντικειμενικός λόγος που να λέμε ότι έχει παραβιαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Ακούμε όλα τα μέρη, αλλά αντικειμενικά και νομικά όχι. Διότι οι αναφέροντες ε, ε, λένε ότι η κυβέρνηση της Καστήλης, η προηγούμενη διοίκηση ενέκρινε το Μάρτιο του 2015, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης που καλύπτει νομικά τις ενισχύσεις που ζητούν, ήταν έξι μήνες αργότερα, 30 Οκτωβρίου 2015. Πώς μπορεί κανείς να λέει ότι παραβιάστηκε ε, ένα πρόγραμμα που δεν εγκρίθηκε η προκήρυξή του παρά έξι μήνες αργότερα. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια πολιτική τσάπα τσουλιά ε, άνευ Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη που υποβάλλει η Μαρία Ντολόρε Ντεκοσπεδάλ, Περιφερειάρχης, το 2013 ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το λαμβάνει αυτό το καλοκαίρι του 2014 έχει πάνω από 67 σελίδες ε, ισχυρισμών. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι τσαπατζούλια και δεν μπορούσε να εγκρίνει αυτό το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης γιατί ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Μόλι θα είπε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικά της λόγια παραθέτω. Ε, ακόμα και έτσι, η κυβέρνηση της Μαρίας Ντολόρες Δέκος δεν λαμβάνει υπόψη αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προκυρήσει βοηθεία το Μάρτιο του 2015, ενισχύσεις δηλαδή, για υποβολή αιτήσεων ε, και δημιουργεί φρούδες ελπίδες για ε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα. Άρα η αναφορά αναφέρεται σε κάτι το προσωρινό ε, που ήταν υπό την αίρεση της ε, τελική έγκριση. Πώ μπορεί να προκηρύξει ενισχύσει, να δημιουργήσεις προσδοκίες στους ε, καλλιεργητέ, χωρί να έχει εγκριθεί το πρόγραμμά σου από εκείνον που είναι αρμόδιο που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την τζαπατσουλιά, τη διοικητική θα πρέπει να διερευνήσουμε. Και αν υπάρχει πρόβλημα να καλέσουμε την Περιφερειάρχη και την κυρία Σοριάνο, την Υπουργό Γεωργία τη περιφέρεια, για να δούμε ότι δύο μήνε πριν τι εκλογέ προκυρίσουν ενισχύσει στον αέρα τελείως, χωρίς να, ε, να έχουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολιτικά και νομικά θεμέλια. 63 σελίδες. Εκεί στην Καστήλη Λαμάντσα γίνεται συζήτηση και αν θα πρέπει να προσφύγουν, να το παραπέμψουν στον Ισαγγελέα την προηγούμενη κυβέρνηση τη περιφέρεια. Πώ είναι δυνατόν να προκυρήσει κρατικές κρατικέ ενισχύσει χωρί να σου έχουν εγκρίνει επίσημα το πρόγραμμα. Άρα, νομικά δεν ευσταθεί αυτό, δεν υπάρχει αντικείμενο, γιατί όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί αντικειμενικά να δημιουργεί προσδοκίε με μια προκήρυξη που δεν ε, πατάει στα πόδια της. Αλλά υπάρχει μια τεράστια πολιτική τσαπατσούλια δύο μήνες πριν τι εκλογέ. Για λόγους προεκλογικούς η κυβέρνηση της Μαρία Δολόρες Δεκοφπεντά ε, αν μη τι άλλο παραπλάνησε τους καλλιεργητές. De, de petición, sujetas... Άρα, δεν υπάρχει θέμα ευρωπαϊκού δικαίου γιατί δεν παραβιάστηκε το πρόγραμμα των ενισχύσεων, γιατί δεν εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αν όμως αποφασίσετε να παραμείνει ανοιχτή η παρούσα αναφορά, προφανώς θα ήταν ενδιαφέρον να διαρευνήσουμε για ποιους λόγους η τότε κυβέρνηση της περιφέρειας προκήρυξε αυτή την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες και να πω το εξή, κοιτάξτε να δείτε. Όταν μια κυβέρνηση εκδίδει μια πράξη, μίλησε ο συνάδελφο Σέρχιο για τη Μαρία Δολόρε στην Κοσπεδάλη. Εγώ δεν θα μπω σε αυτά τα πολιτικά χωράφια. Δεν σκόπευα να το κάνω, αλλά αφού το έκανε ο συνάδελφο, θα το κάνω κι εγώ είναι η Περιφερειάρχης και ο Υπουργός Οικονομίας και ποντάρει στη βιολογική γεωργία. Και εμένα αυτό μου φαίνεται καλό. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω, είμαι σίγουρη. Και βγάζει μια προκήρυξη, ένα διάταγμα που λέει «Ελάτε όλοι και κυβερνήσεις είναι ε, ε, στην υπηρεσία όλων των πολιτών και εκείνους που τους ψήφισαν και εκείνους που δεν τους ψήφισαν». Και έρχεται η επόμενη κυβέρνηση και αρκεί να κάνει κάποιο κάτι έτσι ώστε η επόμενη κυβέρνηση που είναι από άλλο κόμμα να περικόψει. Μα δεν μπορεί να περικόψει αν είσαι βάρο των πολιτών αυτή τη περιφέρεια. Με την περικοπή αυτή, ο κύριο Εμιλιάνο Γκαρθία Πάχε, που τη διαδέχτηκε την Περιφερειάρχη, άφησε ξεβράκο τους και ζητώ συγγνώμη για την έκφρασή μου όλους εκείνους τους καλλιεργητές που αποφάσισαν ε, να ε, προσφύγουν σε αυτές τις βοήθειες. Δύο χρόνια καλλιεργούσαν βιολογικά, είχαν κάποιες προοπτικές εμπορικές, οι οποίες ε, πήγαν στο βρόντο και χάσανε και πάρα πολλά χρήματα από τη βιολογική γεωργία, η οποία δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ενισχύσεις. Οπότε ο πολίτη τι να κάνει, σου λέει τώρα κάνει κάτι η κυβέρνηση, αλλά η επόμενη που θα βγει το άλλο κόμμα θα το ανατρέψει. Είναι αυτό κατάσταση. Και επίση είπαν και αναφέροντε ότι διαταράχθηκε και ε, διαρρήχθη η ε, αρχή τη καλή πίστη και τη αξιοπιστία και τη ασφάλεια δικαίου. Καλό κυβερνήτη είναι εκείνο που διατηρεί τι ενισχύσει, ιδιαίτερα όταν είναι υπέρ του λαού του. Και δεν τις περικόπτει κατηγορώντας τους προηγούμενους που τις υιοθέτησαν. Ας έρθει όποιος θέλει, αλλά να μας εξηγήσει γιατί μια κυβέρνηση της περιφέρειας Καστήλης Δαμάντσα αφήνει πολλούς πολίτες να χάνουν εκατομμύρια από τη βιολογική γεωργία. Το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης βεβαίως έπρεπε να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευρωπαϊκή ε, αρμοδιότητα όμως και ασφαλεία δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή της καλής πίστης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Σβάιτς. Ähm, Ευχαριστώ, θα μιλήσω γερμανικά. Μου είναι πιο εύκολο στο συγκεκριμένο. Καταρχάς θα πρέπει να ε, θέσουμε το εξή ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μια περιφερειακή κυβέρνηση να κάνει περικοπές στη βιολογική γεωργία όταν ο βιολογικός αγρότης με τρόπο υποδειγματικό σέβεται ε, όλες τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Επειδή δεν ξέρω καλά την εσωτερική ισπανική πολιτική, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι που έχει σχέση γενικά για τη γεωργία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και το έχετε αντιληφθεί, αλλά... Όταν οι συμβάσει, οι αγρότε υπογράφουν συμβάσει, αγρότε και αγρότησε μαζί μα, εμεί έχουμε συμβατική υποχρέωση ενοχική να το τηρήσουμε και μάλιστα για όλη την περίοδο. Πενταετία, πενταετία, επταετία, επταετία, αυτά που λέει η σύμβαση. Ποιο είναι το περίεργο. Οι εταίροι μα δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τη σύμβαση. Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τον αγρότη που είναι εκτεθειμένο στην ενίσχυση. Αυτό δηλαδή πρέπει να τα τηρεί, αλλά η άλλη αρχή όχι. Και εδώ βλέπουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι μπορεί να πάθει αγρότη, αγρότησα ή συνεταιρισμό όταν αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και οι πλειοψηφίε. Εγώ θα πρέπει ω αγρότη να τηρώ τη σύμβασή μου, αλλά θα πάρω και τι μισέ ενισχύσει. Και είναι κρίμα. Στην Ευρώπη η γεωργία δυστυχώς εξαρτάται από τις δημόσιες ενισχύσεις για την ίδια της την επιβίωση. Και αυτό ε, πολλές φορές έχει να κάνει με τη ζωή ή το θάνατο μιας εκμετάλλευσης. Για άλλη μια φορά βλέπουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό θέλω να παραμείνει ανοιχτή συγκεκριμένη αναφορά. Peter Κοιτάξτε, υποστηρίζω 100% τον προλαλήσαντα και θέλω να πω το εξή. Πρόκειται για την ίδια την αξιοπιστία και πολύ ωραία τα περιέγραψε. Όταν τελειώνει μια προγραμματική περίοδος και μπαίνουμε σε μια άλλη, ε, υπάρχει μια παροιμία που λέει καινούριο παιχνίδι, καινούρια τύχη. Ε, αλλά δεν μπορείς στα μέσα του παιχνιδιού να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Γι' αυτό θέλω να παραμείνει ανοιχτή αναφορά κι εγώ και τα λέω αυτά από πλευράς και από τη σκοπιά του αγρότη. Ο αγρότη δεν νοιάζεται αν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα ή όχι. Τι τον νοιάζει τον αγρότη, δεν δίνει δεκάρα. Ε, του, του έχουν πει κάνει αίτηση, κάνει αίτηση, κάνει business plan, κάνει τον προγραμματισμό του, κανονίζει την πορεία του. Τι τον νοιάζει ε, ποιο έχει εγκρίνει και τι έχει εγκρίνει γιατί κάνει και άλλε συμβάσει και υπογράφει ας πούμε για την ε, παραλαβή του βιολογικού υλικού και τα λοιπά. Και στη Γερμανία είναι περιφερειακή διάρθρωση, είναι ομοσπονδιακό το, το, κράτος, αλλά δεν ξέρω καμία περίπτωση που να έχει κοπεί, να περικοπεί ένα πρόγραμμα στα μέσα του προγράμματος. Το αφήνουν να τελειώσει, να εκπαιρνεύσει και μετά το επόμενο το κόβουν. Ελάτε λίγο λοιπόν στη θέση των γεωργών, αυτό κοιτάει τι του έχουν βάλει στην τράπεζα το έμβασμα και κανονίσει την πορεία του. Και είναι και ανετική διαφήμιση, είναι δυσφήμιση ουσιαστικά πάρα πολύ μεγάλη. Και μπορούμε να διαπληκτιστούμε πόσα κονδύλια χρειαζόμαστε, αλλά αυτό είναι πραγματικά δυσφήμιση για την Ευρώπη. Και για τη ε, βιολογική γεωργία. Γιατί σου λέει ο αγρότης δεν πάει στο καλό και η βιολογική γεωργία. Ε, νομικά τώρα δεν κατάλαβα, είναι παράνομο αυτό που κάνανε, η περικοπή ε, των ενισχύσεων. Μπορούσαν να το κάνουν, επιτρεπότανε. Βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Και ως αγρότης εγώ θα έκανα και ε, διαδήλωση και θα πήγαινα να ξεφορτώσω το, την παραγωγή μου καλά καλά. Δεν θέλω να το τραβήξω, ξέρω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν αγρότης. Ε, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ε, αξιοπρεπής και ευπρεπής ε, απέναντι στον επαγγελματικό κόσμο και τον αγροτικό κυβερνήση. Ο κύριος Τερικά Μπράς. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα από τους συναδέλφους. Συμφωνώ. Αυτό που θα επιθυμούσα είναι σε τέτοιες συζητήσεις να είχαμε περισσότερη λογική να πριτανεύει και λιγότερο κομματική λογική. Να ε, μην θέλει ο ένας να την μπαίνει στον άλλον. Εδώ ακούσαμε ότι ε, ελήφθησαν μέτρα με αναδρομική ισχύ. Και αυτοί οι ίδιοι που διαμαρτύρονται τώρα έχουν λάβει αναδρομικά μέτρα για την ενίσχυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπήρχαν ενισχύσεις για τις ΑΠΕ και έχουν λάβει μέτρα αναδρομικά για να τα καταργήσουν. Πραγματικά πολύ θεαματικά και πολύ αντιευρωπαϊκά πράγματα. Αλλά σας λέω, ε, μην μπαίνουμε σε αυτή τη μικροψυχία τώρα της κομματικής συζήτησης και της μικροκομματικής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, αντικειμενικά κριτήρια, ανάληψη ευθυνών ε, και τήρηση των ε, υποσχέσεων. Βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να την ψάξουμε σε βάθος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε εκ νέου τώρα στους αναφέροντε. Παρακολουθήστε την όλη συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Ακούσατε επίση ε, την παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε λοιπόν το λόγο για δύο λεπτά ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω λίγο ε, να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Σάρχιο Γκουτιέρεθ, που είναι και συντοπίτη μου. Εμείς είμαστε γεωργοί. Υπογράψαμε μια σύμβαση που μας έφερε η διοίκηση με τις δικούς τους όρους. Εμείς ούτε όρους βάλαμε, ούτε χρόνους βάλαμε. Και ε, εκείνοι παραβιάζουν τη σύμβαση. Και αν δεν έχουν χρήματα να αλλάξουν τις ποσοστώσεις, να αλλάξουν ε, τις συνθήκες και αυτός που θέλει να συνεχίσει να είναι βιολογικός γεωργός να συνεχίσει. Αλλά τη σύμβαση θα πρέπει να την τηρήσουν. Αλλιώς δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου συνοψίζω λίγο αυτά που άκουσα πρώτον. Θέλω να πω ότι ε, κάναμε μια συζήτηση στο ΛΕΔΟ με, το Φιλ ε, Χόγκαν και ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας ε, αναγνώρισε ότι μπορεί να κάνανε και λάθος. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι έσφαλες, αλλά πρέπει να διορθώσεις και το λάθος σου. Σε ό,τι αφορά την ανασταλτική ρήτρα, είπε ότι δεν μπορούσανε ε, να ανακοινώσουν ε, τις ενισχύσεις ε, εφόσον εκκρεμούσε η έγκριση του σχεδίου. Όλοι είχαμε καταλάβει ότι αν δεν εγκριθεί το σχέδιο δεν θα ερχόντουσαν λεφτά. Αλλά εάν εγκρινόταν από την Ευρώπη θα παίρναμε αυτά που μας είχαν τάξει, όχι ότι θα αλλάζανε τα ποσά στη μέση του δρόμου. Σε αρχαίο μπορεί να σου φαίνεται ε, τσαπατσουλιά ή όχι, αλλά το έχει χρησιμοποιήσει και ο Μπόνο και ο Μπαρέρα και ο Γκαρσιαβάσκε, δηλαδή διάφοροι περιφερειάρχες διαφόρων κομμάτων δεν μπορεί να αλλάζει η ερμηνεία κατά το δοκούν ανάλογα με τον Περιφερειάρχη. Ο καθένας όπως θέλει. Και ακούσαμε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προκήρυξη και το σχέδιο και ότι όλα ήταν σύνομα. Και το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης είχε ε, υπολογισμούς για τις ποσότητες, για τις ζημίες και τα λοιπά. Ξέραν τι χάνουμε και πού βρισκόμαστε. Και σε σχέση με το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώς η Καστήλη Λαμάντσα δεν είναι πολύ παραγωγική περιφέρεια και είναι μεγαλύτερες οι απώλειες. Δεν είναι πολύ γόνιμη η γη. Και πάντα χρειάζεται την ίδια φροντίδα στη βιολογική καλλιέργεια, ανεξαρτήτως της παραγωγής, των ποσοτήτων δηλαδή και για τις επιφάνειες 365.000 εκτάρια ήταν το 2015. Από την αρχή ήταν γνωστές οι επιφάνειες. Τώρα, αν δεν ε, διορθώσει το σφάλμα της η περιφέρεια της Καστέλης Λαμάντσα, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη βιολογική καλλιέργεια κάποιοι γεωργοί, γιατί δεν είναι ε, αποδοτική η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική ως προς τη γεωγραφία και θα υπάρξουν ε, περιφέρειες που δίνουν περισσότερο ποσοστό στην βιολογική καλλιέργεια, άλλες λιγότερο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει μια αυτόνομη περιφέρεια να παραβιάζει την ασφάλεια δικαίου. Και όπως ακούστηκε επανειλημμένα, η σύμβαση είναι κάτι το οποίο θεσμεύει και θα πρέπει να τηρήσεις την υπογραφή σου. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ που ήρθατε εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες για να μας παρουσιάσετε την πολύ πολύπλοκη αυτή αναφορά, ιδιαίτερα πολύπλοκη και για πολλούς και διάφορους λόγους και βέβαια και για πολιτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο στην αφορά αυτή από πέρυσι το καλοκαίρι. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Δεν υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία σε αυτή την αναφορά, Ωστόσο όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολιτικά ευαίσθητο. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να το διερευνήσουμε λίγο περισσότερο και συνεπώς σας προτείνω αυτό βλέπω ότι θέλουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι. Εγώ θα μπορούσα να προτείνω κάτι διαφορετικό. Προτείνω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να αποσταλεί μάλιστα και στην Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου και να του ζητήσουμε να γνωμοδοτήσουν για αυτή την αναφορά. Ξέρετε ότι από νομική πλευρά εμπίπτει σαφώ στην αρμοδιότητα τη Επιτροπής Γεωργία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τους αποστείλουμε όχι μόνο μια επιστολή ενημερωτική, αλλά να τους ζητήσουμε να εκπονήσουν και μια γνωμοδότηση, να διερευνήσουν περισσότερο το ζήτημα και να μας πούνε τελικά αν τα όσα έχουν συμβεί στην περιοχή αυτή συνάδουν με την ανοσιακή νομοθεσία. Και βλέπω ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι ε, πρέπει να αποχωρήσω γιατί θα πάω στο Brexit Steering Group. Και θα έχετε τώρα τη χαρά να έχετε έναν πολύ καλύτερο πρόεδρο, τον Πολ Τσάλκι. Πρέπει λοιπόν να πάω στην άλλη συνεδρίαση. Δεν νομίζω ότι θα, θα για πάρα πολλή ώρα. Πάντως με τον Πάτη είστε σε πάρα πολύ καλά χέρια. So, gentlemen, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, Ουγγρικά λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισσιας διαταξης διάταξης, αναφορά 15-25 2016, ένα ζήτημα ιδιαίτερα πολύπλοκο και ιδιαίτερα ευαίσθητο κιόλας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αριάσα, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν 379 υποθέσεις ανεξιχνίας των επί του παρόντος δολοφονιών που έχουν διαπραχθεί κατά πάσα πιθανότητα από την τρομοκρατική ομάδα ΕΤΑ στην Ισπανία. Τον Οκτώβριο του 2017, στις 11 Οκτωβρίου του 2017, κάναμε μια πρώτη συζήτηση για αυτή την αφορά στα πλαίσια της Επιτροπής μας και στη συνέχεια αποφασίσαμε ότι το ζήτημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και ευαίσθητο και είπαμε ότι θα έπρεπε να αποσταλεί μια επιστολή προς την Ισπανική κυβέρνηση και επίσης ζητήσαμε τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα διαβήματα, να σημειώσουμε πρόοδο. Το θέμα τώρα είναι ότι λάβαμε απαντήσεις σε ορισμένες μόνο από τις, από επιστολές που στείλαμε. Από ό,τι φαίνεται όμως η Επιτροπή Αναφορών δεν είναι ικανοποιημένη με την ποιότητα των απαντήσεων αυτό και γι' αυτό το λόγο ορισμένοι συνάδελφοι ζήτησαν από την Επιτροπή μας να διεξαχθεί μια δεύτερη συζήτηση για αυτή την αναφορά και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας δώσω τώρα το λόγο. Θα ήθελα όμως καταρχάς να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των αφέροντα, δηλαδή είτε στον Ντάνιελ Πορτέρο τώρα ή στον Μιχέλ Άγχελ Ροντρίγκερς Αρίας. Έχετε το λόγο συνολικά για πέντε λεπτά. Γεια σας. Καλησπέρα σας σε όλους και σε ευχαριστούμε πολύ που μας ε, δέχεστε. Θέλω να θυμίσω ποιος είμαι. Πρόεδρος μιας οργάνωσης αλλά και γιος ενός δολοφονηθέντος από την ΕΤΑ, από τους 856 που δολοφόνησε αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Ο πατέρας μου ήταν δικαστής στην Ανδαλουσία, επικεφαλής κιόλα δικαστής και εδώ δεν είμαι μόνο εγώ παρόν, έχουμε και άλλους συγγενείς δολοφονηθέντων. Η Μάιτε Παγάσα Ορτοντούα, η Τερέσα Χιμένεθ Μπεχερέλ που έχασαν μέλη της οικογένειάς τους που δολοφονήθηκαν. Από κοινού έχουμε ένα κοινό στόχο μάλλον ο στόχος της ΕΤΑ ήταν να αποσταθεροποιήσει ε, ε, το κράτος. Στο πατέρα μου ήταν εισαγγελέα. Ε, στην Τερέσα Χιμένεθ Μετερή, ο αδελφός της Μάιτε Παγάσα και ε, της Τερέσα Χιμένες ήταν στις ε, δυνάμεις ασφαλείας. Και το πρόβλημα ποιο είναι από τους 856 φόνους στις δολοφονίες, 379, περίπου 400 δεν έχουν εξηχνιαστεί. Δεν έχει προχωρήσει η Ισπανική αστυνομία και δικαιοσύνη. Όπως είπατε, αντιλάγησαν επιστολές, απάντησε η εισαγγελία της ε, Audiência Nacional, που είναι το ειδικό δικαστήριο, υπουργό δικαιοσύνη, με κάποιες ασαφείς και αφηρημένες και πολύ γενικές παρατηρήσεις και έλεγε ότι φταίει η δικαιοσύνη, η Audiencia νασιονάλ το ειδικό δικαστήριο. Η εισαγγελία της ε, Audiencia νασιονάλ έστειλε μια έκθεση του 2011 μετά από αναφορά ε, της τότε Προέδρου ε, της Ένωσης των Θυμάτων που είναι τώρα ε, προβουλευτής και εδώ παρούσα η Μαϊτέ Παγάσα Ορτοντούα αλλά από το 2011 και 2017 δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει ενημερωθεί τίποτα. Δύο στις τέσσερις απαντήσεις είναι απολύτως ασαφείς και γενικόλογες και κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης εστάλει ε, επιστολή στον πρόεδρο του ειδικού δικαστηρίου που δεν έχει απαντήσει και απομένει η Ντολόρης Δελγάδο που είναι πολύ ειδική εισαγγελέα και πολλοί εμπειρογνώμων που ε, έχει λάβει την επιστολή αλλά δεν απάντησε και θα πρέπει να την ξαναστείλετε. Και μάλιστα τώρα μόλις η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας την όρισε, τη διόρισε Υπουργό Δικαιοσύνης. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να της ξαναστείλετε αυτή την επιστολή στην κυρία Ντολόρες Ντελγκάδο που ήδη είχατε κάνει. Επίσης, επειδή δεν έχει απαντήσει καθόλου ε, η Ισπανία να ζητήσετε από την ε, Ισπανική αστυνομία, χωροφυλακή, ε, υπηρεσίε πληροφοριών και από τον ίδιο το συνήγορο του πολίτη που τόσο έχει ψάξει ε, σε αυτέ τι ανεξιχνίαστε περιπτώσει. Υπάρχουν θεσμοί, όπω είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ισπανία, που θα είχε να σα πει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Αλλά το σημαντικότερο και επιμένω είναι ότι θέλουμε να ε, μεταβεί αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί ακριβώς σε αυτούς τους θεσμούς και να ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έχουν διερευνηθεί αυτά. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ είμαι εγώ η φωνή πολλών θυμάτων της τρομοκρατίας. Και έχω αυτή την κληρονομιά σήμερα. Αυτούς εκπροσωπώ. Όλους εκείνους που σήμερα πια δεν έχουν φωνή εδώ. Τον ίδιο τον πατέρα. Ο πατέρας μου δικαιώθηκε. Αλλά περίπου οι μισοί δεν έχουν δικαιωθεί από τα θύματα. Έχουμε απαντήσει ότι η Ισπανία επανόρθωσε. Τι, τίποτα δεν επανόρθωσε. Και το χειρότερο, στο χειρότερο θέλω να εστιάσω. Μας είπαν ψέματα από την Αουδιένθια Nacional που είναι το μεγαλύτερο ειδικό δικαστήριο στην Ισπανία ε, ε, που δικάζει ε, θέματα τρομοκρατίας. Και το λέω ξεκάθαρα εδώ. Ψεύδι ήταν αυτά που μα είπαν και το λέω γιατί έχουμε προσφύγει εκεί από τους 379 έχουν δύο περιπτώσεις, τον Μανουέλ Θαμαρένιο, δημοτικός σύμβουλος του Παρτίδο Ποπουλά στην Κυπούθκουα και ο Χωσέ Λουίς Κάσο που έξι μήνες αργότερα τον διαδέχθηκε. Όχι, πρώτα ήταν ο Χωσέ Λουίς και μετά ο Μανουέλ. Και οι δύο δολοφονήθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν δημοτική σύμβουλη του Λαϊκού Κόμματος του Ισπανικού και συστηματικά τους δολοφονούσε η ΕΤΑ. Και το χειρότερο είναι ότι το ίδιο αυτό το δικαστήριο, Αντιένθια Ναθιονάλ, έφτασε να πει πριν από δύο εβδομάδε ότι η συμπεριφορά των δύο αυτών κυρίων ήδη έχουν ε, τιμωρηθεί οι δολοφόνοι. Α, μας λένε ότι πλήρωσαν δηλαδή. Το έκτο τμήμα του δικαστηρίου στις 14 Φεβρουαρίου 2018 ε, σε έτους ότι έχουν τιμωρηθεί αυτοί οι, οι και με σχετική έκθεση που έρχεται να αντικρούσει άλλες εκθέσεις. Παρακαλώ διαβάστε τι σας έστειλε εισαγγελία που λέει ότι αυτοί οι δύο κύριοι ε, είναι δύο περιπτώσεις που δεν έχουν εξυχνιαστεί. Ε, το λέει στη σελίδα νέα της έκθεσης που έστειλε ο εισαγγελέας και το έχετε στα χέρια σας. 15 Πρώτου 2017 η ημερομηνία και στη σελίδα 25 της ίδιας έκθεσης που λέγουν ότι δεν έχουν βρεθεί η αυτοργοί, ότι ε, δεν έχουν λυθεί. Ενώ στο παρελθόν μας έχουν πει ότι τιμωρήθηκαν οι ένοχοι. Δεν θέλουν να ε, εξεχνιάσουν τις μισές περιπτώσεις δολοφονιών και ψεύδονται και το λέω έτσι ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια και επιμένει πάρα πολύ η International να χρησιμοποιεί αυτά τα δύο παραδείγματα, τις δύο περιπτώσεις ω σαφή παραδείγματα. Και εμεί έχουμε ενδείξει ότι δεν ε, έχουν καθόλου την πρόθεση να τα λύσουν αυτά, να τα εξηχνιάσουν. Και λέει το κατηγορητήριο ότι όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση ΕΤΑ ήταν αντικείμενο αστυνομικής και δικαστικής διερεύνησης. Αυτό το λέει το ανώτατο αρμόδιο δικαστήριο. Και έχουν δικαστεί είτε στην Ισπανία είτε στη Γαλλία. Και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συλληφθεί, απαγγελθεί κατηγορίες, κατηγορηθεί και καταδικαστεί η υπέτειοι όλων αυτών των εγκλημάτων. Ψεύδονται και λένε όσοι έχουν αναγνωριστεί ως θύματα της ΣΕΤΑ έχουν λάβει επανορθώσεις και αποζημιώσεις ακόμα και όταν δεν ε, ταυτοποιήθηκε ο, ο ε, ένοχος. Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν ε, ρυθμίσεις και νομοθεσία. Ψεύδονται από το 1999 Ούτε δύο δεκαετίε δεν έχουν περάσει. Όταν λένε πολλέ δεκαετίε στον πληθυντικό, τουλάχιστον θα πρέπει να περιμένει να περάσει και η δεύτερη δεκαετία να ολοκληρωθεί. Και λέω ότι ψεύδονται γιατί όλα τα εγκλήματα δεν έγιναν. Από τους 379 υπάρχουν 7 περιπτώσεις ε, εξολόθρευσης μάλλον ε, ε, που έχουν χαθεί όλα τα στοιχεία ε, τον από τα αρχεία, έχουν εξαφανιστεί οι δικογραφίες και δεν μπορούν να τα διερευνήσουν. Πάνω από 200 περιπτώσεις από τις 379 δεν φτάνουν τα 100 φύλλα, 100 σελίδες δηλαδή και το χειρότερο πάλι από το Δικαστήριο Αντιένθια Ναθιονάλ, γι' αυτό επιμένω που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Αναλύεται η κατάσταση μόνο από το 1978 και μετά. Η ΕΤΑ συστήθηκε το 1959 και οι εκθέσεις που έχει στείλει το Δικαστήριο Αντιένθια Ναθιονάλ είναι από το 1978 και μετά. Για ποιο λόγο? διότι φοβούνται τον περίφημο νόμο αμνηστίας που ήρθε το 1977. Δηλαδή αν πήραν το 77 αμνηστία οι δολοφόνοι, έχουν αμνηστία και τα θύματα. Δηλαδή πήραν αμνηστία και τα θύματα, ότι δεν έχει δικαίωμα να δικαιωθεί τώρα, να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έχει υπέρθει αμνηστία και αυτό είναι ε, ακατανόητο, διότι από το 1959 μέχρι το 1977 είχαμε 70 ανεξιχνίαστες υποθέσεις, που αν προσθεθούν σε όλες τις υπόλοιπες σχεδόν φτάνουν στις 400 που είναι μισές. Δεν το έχει διερευνήσει λοιπόν το δικαστήριο αυτό. Ε, ε, δεν έχουν ψάξει ε, τους ηθικούς αυτοργούς, ε, τους εντολοδόχους, τους ε, ηγέτες. Πάντα ψάχνουν περίστροφα, συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίοδο των Ναζί υπήρξαν στοιχεία που μπόρεσαν να βοηθήσουν να καταδικαστούν οι ηγέτες και εκείνοι που έδιναν τις εντολές και κινούσαν τα νήματα. Έχουμε πάρα πολλά εμπόδια και φραγμούς στην διερεύνηση ε, αυτών των πραγμάτων και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παρόλο που το έχει αναγνωρίσει αυτό η Ισπανία και από το 2004 εφαρμόζεται, χρειάστηκε να πάμε στην Αργεντινή για να ε, διερευνηθούν οι περιπτώσεις πριν από το 2014. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σας παρακαλώ, στείλτε λοιπόν αντιπροσωπεία. Σας παρακαλώ, ζητήστε περισσότερες εκθέσεις και από άλλους θεσμούς, από την αστυνομία, από την Αντιένθια Νασιονάλ, αλλά ουσιαστικά αισθανόμαστε ανυπεράσπιστοι και απροστάτευτοι. Από τη δικαιοσύνη θέλουμε να αποζημιωθούμε, δεν θέλουμε χρήματα, μόνο δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε την ε, κυρία Πλούμσπαρ που θα μα εκθέσει την άποψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το ζήτημα είναι ευαίσθητο. Και θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα εκφράζοντας και εγώ την ε, υποστήριξή μου και ε, την, προς τους ετούντες και προς τα, όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Όμως, οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προκειμένου είναι περιορισμένε και είναι λίγα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τι συγκεκριμένε εγκληματικέ πράξει. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να βοηθήσουμε τα θύματα τη δημοκρατία συνολικά. Το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Έχουμε πλέον ψηφίσει οδηγία η οποία θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη χρονιά όσον αφορά την υποστήριξη των θυμάτων τη τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και τη ε, ε, υποστήριξή τους της οικονομικής μετά της αναγνώρισης του στάτους του θύματος. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες είτε από το 2018 είτε αμέσως μετά. Θα δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού για τα θύματα της ένοπλης βίας στην Ευρώπη, στην Και βέβαια θα γνωρίζετε ότι υπάρχει και ο ειδικό σύμβουλος του Προέδρου της Επιτροπής ε, που θα του υποβάλει προτάσεις για την υποστήριξη και ε, την βοήθεια προς τα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτά οι πρωτοβουλίες είναι ε, σωστές και φταίες και πολύ καλές, αλλά βεβαίως δεν σας βοηθούν εσάς και δεν σας αποδίδουν δικαιοσύνη στις δικές σας υποθέσεις. Όμως είναι το μόνο που μπορώ να πω ως προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουμε την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στο μέλλον. Ο Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Κυρία Σταράς Φαραγκούτ, ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες και όλος ιδιαίτερος τη Μάιτα Παγάσα Ορτουντούα και την Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλ που εκείνες μαζί με εσάς ε, είναι οι πλέον ενδεδειγμένες να καταδείξουν και να αναδείξουν το πρόβλημα. Στις 11 Οκτωβρίου είχαμε μια συνεδρίαση πολύ συγκινητική και πάρα πολύ φορτισμένη. Πάνω από 44% των ε, εγκλημάτων δεν έχουν ε, ξεχνιαστεί και δεν είναι εύκολο για κανένα και παραγράφονται κιόλας ε, αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει μια ολόκληρη οργάνωση από πίσω και η τελευταία δολοφονία έγινε στη Μαγιόρκα την πατρίδα μου και δεν έχουν καταδικαστεί οι ε, χωροφύλακες ε, αυτοί που δολοφονήθηκαν και σε λίγο παραγράφεται το έγκλημα. Οι απαντήσεις δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων της, ε, του αιτήματό μας και της αναφοράς σας. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπαν οι αναφέροντες. Θα ακούσουμε τις συναδέλφους Μάιτε και Τερέσα και τους υπολείπους, τους Ζεπ, και όποιος θέλει να μιλήσει. Αλλά Σύμφωνο να απευθυνθούμε στις δυνάμεις ασφαλείας, ε, στην αστυνομία, στην χωροφυλακή, τις μυστικές υπηρεσίες, στο συνήγορο του πολίτη, στην Ντολόρες Δελγάδο, στο Υπουργείο ε, Εσωτερικών και να στείλουμε και αποστολή. Μακάρι να μπορούσαμε κατά προτεραιότητα να πάμε στην Ισπανία. Το Σεπτέμβριο έχουμε μια επίσκεψη, μια αντιπροσωπεία στην Τονιάνα που είναι ο δρυμός αυτός στην Ισπανία, το Εθνικό Πάρκο, αλλά και τούτη εδώ είναι προτεραιότητα. Μετά θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο, αλλά θα ζητήσω από τον Προεδρεύοντα τώρα και την Πρόεδρο της Επιτροπής να μην τα αφήσουν αυτό στη τύχη του, να ε, εγκριθεί η αποστολή. Ελπίζω να το εγκρίνουν οι συντονιστές. Η Κομισιόν μας λέει ότι το κράτος μέλος είναι αρμόδιο. Ζήσαμε πολλές περιπτώσεις όπου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει αρμοδιότητες, όπως η περίπτωση της απαγωγής των παιδιών, των απαγωγών αυτών, ε, που, τηρουμένων των αναλογιών. Αλλά χρειάζεται ε, επίσκεψη. Πήγαμε στο Γενικό Εισαγγελέα, στις δικαστικές αρχές, στο Υπουργείο, γιατί και η δική μας Επιτροπή χρησιμεύει στο να αφυπνίζει συνειδήσεις και να αφυπνίζει και θέματα που ε, κοιμούνται και να δημιουργεί αντιδράσεις θα το διαβιβάσω στο συντονιστή μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία. Και σας στηρίζω πώ αλλιώ άλλωστε θα γινόταν αλίμονο όλες τις οργανώσεις και όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεχνιαστούν αυτές οι περιπτώσεις που είναι πάνω από 44% και είναι και πολύ ανισχυτικό γιατί πολλές φορές φαίνεται ότι δεν ε, έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Για να δούμε. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε ω Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τερέσα Χιμένε Μπεσερίλ. Τερέσα να με λέτε, γιατί το επίθετο είναι δύσκολο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Έχω την τύχη να γνωρίζω ποιος σκότωσε τον αδελφό μου, ποιος τον δολοφόνησε, Αλμπέρτο Χιμένες Μπεσερίλ, ε, αντιδήμαρχος της Σεβίλη ήτανε, 36 χρονών και τη γυναίκα των Σεσιών Γκαρθία Ορτής. Έχω αυτή την τύχη. Λίγες εβδομάδες μετά τους συνέλαβαν και τώρα εκτείουν την ποινή τους από το 99 σε μια φυλακή στην Ισπανία. Αλλά οι οικογένειες του Χουάν Μανουέλ, του Αντώνιο, του Ντιέγκο, του της Χωσεφίνα, της Μαργαρίτα και άλλων πολλών δεν έχουν την τύχη που είχα εγώ ή την τύχη που είχε η Μάιτε ή ο Ντάνι που γνωρίζουμε ποιος σκότωσε τους συγγενείς μας. Εκείνοι δεν γνωρίζουν ούτε ποιος ε, τράβηξε τη σκανδάλη, ε, ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος το αποφάσισε, ούτε καν και σημαντικότερο, το σημαντικότερο, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Ντάνι και η Μάιτε για μας, ποιος διέταξε τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων. Καμιά φορά είναι δύσκολο να βρούμε τους φυσικούς αυτοργούς, αλλά ξέρουμε ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτούργοι. Αυτούς θα πρέπει να κυνηγήσουμε, γιατί τους γνωρίζουμε ποιοι ήταν. Ε, Άρα η δήλωση που έκανε η ΕΤΑ έτσι, με προπαγανδιστικό τρόπο και τυμπανοκρουσίες, με μια ΕΤΑ η οποία είχε ήδη ιτηθεί που ανακήρυξε ότι διαλύεται, πρέπει να το ξέρετε, αγνόησε ε, ανα πάσα στιγμή τα θύματα. Όταν ζήτησαν συγγνώμη, αυτό το συγγνώμη ήταν μικρόψυχο. Ήταν ένα συγγνώμη που δεν αφορούσε τον αδελφό μου που ήταν πολιτικός, ούτε τη Μάιτε, γιατί ήταν επικεφαλής της Ερτσάντσα, της ε, βασικής Αστυνομία ούτε τον πατέρα του Ντάνι επειδή ήταν εισαγγελέα. Αυτή η συγγνώμη σε ποιον φτάνει, σε κανένα από τα θύματα. Οπότε μην μα κοροϊδεύουν κιόλας. Αυτό το τέλος λοιπόν της ΕΤΑ δεν μπορεί να σημαίνει τελεία και παύλα. Γιατί, ε, Ντάνι, με κάλυψες, δεν έχω να προσθέσω. Σχεδόν 400 εγκλήματα είναι ανεξεχνίαστα και ποτέ εμείς δεν θα ε, δεχτούμε ένα τέρμα ε, στην τιμωρία. Θα πρέπει, ε, θέλουμε να επιβληθεί τέρμα στην ατιμορρησία. Αυτές οι επιστολές, όπως είπε και η Ρώσα, ουσιαστικά δεν μας λένε τίποτα. Άρα θέλουμε να υπάρξει μία συνέχεια σε αυτή την αναφορά, να, κάνουμε κάτι παραπάνω. Έχουμε ξαναζητήσει αποστολή στην Ισπαρία και νομίζω ότι είχε αποφασιστεί και ήταν και πολύ περισσότεροι βουλευτές παρόντε και όλοι συμφώνησαν να γίνει αυτή η αποστολή. Αυτό γιατί σταμάτησε ξέρω ότι δίνεται προτεραιότητα, δίνεται με ΑΙ σε άλλε αποστολές ε, που είναι και αυτό σεβαστό, αλλά σεβαστή είναι, αλλά εδώ δεν καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Είναι εκατοντάδες οικογένειες που απαιτούν δικαιοσύνη και αλήθεια που τους αξίζει. Και η ΕΤΑ ποτέ των ποτών δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Η ΕΤΑ γνωρίζει Ποιο δολοφόνησε, ποιο τον έστειλε, τα πάντα τα ξέρουν. Και τώρα κάνουν αυτή τη δήλωση ε, ε, παράδοση όπλων και τερματισμού. Ε, ήταν υποχρεωμένοι να συνεργαστούν με τη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά ζητούν διάφορα πράγματα, αλλά δεν συνεργάζονται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από την ΕΤΑ, γιατί είναι σκέτη τρομοκράτες και σκέτη δολοφόνοι. Εμεί όμω είμαστε με τη δικαιοσύνη, με την αλήθεια και με τη μνήμη. Και εμεί έχουμε όντω το δικαίωμα να ε, τους δώσουμε στα θύματα και σε όλες τις οικογένειες ένα παράθυρο ελπίδας. Παρακαλώ λοιπόν όχι απλώς να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, αλλά να γίνει και αποστολή στην Ισπανία για να δούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Συνέγορο του Πολίτη, την Υπουργό Δικαιοσύνης τον ε, Γενικό Εισαγγελέα, την ηγεσία της χωροφυλακής και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να μας βοηθήσει. Για αυτή την αφορά μνήμης ε, αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Και θέλω να πω μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, γιατί γνωρίζω όλα αυτά που αναφέρετε και τις οδηγίες και τις γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί έχω συνεισφέρει. Ιδιαίτερα για την οδηγία για τα θύματα την έκανα το 2011 και τώρα παρακολουθώ την εφαρμογή. Ξέρω πάρα πολύ καλά μέχρι που φτάνουν, τι περιλαμβάνουν και τα λοιπά. Τα περισσότερα είναι σε αιτιολογικές σκέψεις και δεν καλύπτουν ε, τα θύματα της τρομοκρατίας. Παρ' όλα αυτά εγώ το παρακολουθώ και ελπίζω ε, και εσείς πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ λίγα τα πράγματα που δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά, ούτε να στηριχθούμε σε αυτά. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τις αρμοδιότητες, αλλά η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και θα πρέπει να την έχει, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, θύματα μη να έχουν ισότητα στο δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό ζητούν τα θύματα και εμείς θα πρέπει να τους το εκχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η Μάιτε Παγάσα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναφέρθηκε ο αδερφός μου. Γι' αυτό θέλω κάτι να διευκρινίσω. Τον δολοφόνησαν επειδή ήταν φυσικός ηγέτης. Ήταν ε, ε, ηγέτης το Σοσιαλιστικό Κόμμα του χώρα των Βάσκων, Εουσκάδικο Εσκέρα και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια ομάδα που ιδρύσαμε, Βάσκοι πολίτες, πήρε το βραβείο Ζαχάροφ το έτος 2000. Το 2003 δύο από τους φίλους μας, ο ένας ήταν αδελφός μου, ο άλλος ήταν ο Χουσέ Λουίς, αντιφραγκιστής, ακτιβιστής, δημοσιογράφος και οι δύο δολοφονήθηκαν. Ομάδα ακτιβιστών που είχε βραβευτεί με το βραβείο Σαχάροφ το 2000. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό το λόγο το δολοφόνησαν και τον κυνηγούσαν. Ξέρετε ότι θα σας φαίνεται πολύ περίεργο. Ε, πώς είναι δυνατόν τέτοια ατιμορρησία συσσωρευμένη, για πολλούς λόγους, όχι ένα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Στη χώρα των Βάσκων, ε, πολύ περισσότερο από τις δολοφονίες ήταν ο εκφοβισμός. Οι δολοφονίες ήταν σταγόνα, ομοιοπαθητικοί μιας ολόκληρης δομής τρόμου και διώξεων, συνδύσεων. Κάτι που θα έμοιαζε περισσότερο με την Ιταλική μαφία ε, σε θέματα ταυτότητας και δολοφονικής πρόθεσης. Διαβάζω τα πρακτικά ε, του γκέτου της Βαρσοβίας και ζω πράγματα που, βλέπω πράγματα που τα έχω ζήσει. Στο οικοσύστημα του τρόμου που ζούμε, που ζούσαμε και χρειάζεται να γίνουμε ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θέλω να σας αναφέρω μία μόνο περίπτωση. Υπήρξε μία περίπτωση δολοφονία στο Σαν Σεβαστιάν και εδώ σε αυτά τα έγγραφα και, και μόνο στο Σαν Σεβαστιάν και στο δικό μου το χωριό το Αλάου είναι πάνω από 30 τα ανεξιχνία στα εγκλήματα. Στο Σαν Σεβαστιάν που είναι από τι πιο, πιο του κόσμου και ε, δημιουργήθηκαν πολλά τραύματα και πολλές ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα, καταστήματα. Και ο, τότε δικαστής που δεν υπήρχε ειδικό δικαστήριο στη Μαδρίτη άφησε ανοιχτή την υπόθεση μέχρι να πληρωθούν οι αποζημιώσει για τι υλικέ ζημίε. Και ακριβώ την επομένη πέταξε στον κάθε των αχρήστων την έκθεσή του. Τι θέλω να σας πω με αυτό, ότι είναι απαραίτητο και για λόγους ηθικής αποζημιώση. Ψυχική οδύνη να πάει αντιπροσωπεία στην Ισπανία, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι πιστεύετε και από ό,τι λένε οι κανόνε. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Ε, μπορούμε να στείλουμε νέε επιστολέ, αφού δεν απαντήθηκαν όλε. Και γιατί υπάρχουν ε, και κάποια σφάλματα στι απαντήσει. Και βεβαίω μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουμε την μετατρομοκρατία εποχή. Και εκτός από τη δικαιοσύνη υπάρχει και η αλήθεια. Και εμεί ω ευρωβουλευτέ, και ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιους να έχουν μια στοιχειώδη ηθική ντροπή με νέα στοιχεία, σε κάποιους που είναι ξαδιάδροποι, ε, με νέα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν. Να το κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Εγώ κανονικά δεν θα έπρεπε να πάρω το λόγο. Είναι τόσο δραματικά τα πράγματα, τόσο τρομακτικά. Εδώ και ώρα έχει αρχίσει άλλη συνεδρίαση που έπρεπε να είμαι παρόν, αλλά δεν θέλησα να φύγω Ακριβώ για να είμαι παρόν και να σας εκφράσω την αγάπη μου, τη συμπόνια μου και τη συλληπιτήριά μου. Είναι πραγματικά ιδιαίτερο η δεχτή όλα αυτά. Θέλω να επιμείνω, συμφωνώ απόλυτα να επιμείνουμε, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται. Το θέμα είναι αστυνομικό και δικαστικό. Αν θέλουν οι συνάδελφοι, συμφωνώ με την αποστολή και την αντιπροσωπεία, αλλά θέλω να θυμίσω επίσης ότι χρειάζεται και διερευνητική ε, αποστολή των πραγμάτων. Μάλλον το fact-finding χρησιμεύει στο να αποκαλυφθούν γεγονότα. Είναι γνωστά τα γεγονότα και είναι και τρομερά. Δεν είναι να πάμε στην Τονιάνα, στο φυσικό δρυμό, να δούμε τι κάνουν και πώς επιδεινώνεται η κατάσταση. Δεν χρειάζεται ερευνητική των πραγμάτων επιτροπή εξεταστική. Είναι γνωστά τα πράγματα, είναι η και ολέθρια. Δεν ξέρω αν χρειάζεται αν θέλετε να μου πείτε πάμε και πάω και με τα πόδια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πού να πάμε και τι να κάνουμε. Και να ε, πιέσουμε σε όλα τα επίπεδα και γράμματα και επιστολές, αιτήματα, ό,τι θέλετε. Εκστρατείες βεβαίως, απολύτως σωστό και ε, επιβεβλημένο. Και μεταξύ άλλων, διότι, και επιτρέψτε μου αυτή τη σκέψη, ακόμα και αν δικαιωθείτε, ποτέ δεν δικαιώνεται κανείς. Δηλαδή, έχουν χαθεί οι άνθρωποι αυτοί. Πόσο πληρώνεται, με 20 χρόνια, με 400 χρόνια κάθερξη. Πώς εξαγοράζεται αυτή η ποινή. Και η τεράστια οδύνη που ζει κανείς δεν ε, απαλύνεται. Θα την, έχετε, ε, θα την έχει κανείς όλη τη ζωή. Τώρα, αν θέλετε να στείλουμε αποστολή και αντιπροσωπεία και θεωρείτε ότι είναι χρήσιμη, Εμπρός, λοιπόν. Αλλά μην νομίζουμε ότι θα κάνουμε και τίποτε επειδή θα πάμε εκεί ή ότι θα τα επιτύχουμε όλα. Εγώ θα υπερψηφίσω. Απλώς θέλω να πω και να εκφράσω την οδύνη μου και τη συντριβή μου ότι θέλω κάτι να γίνει. Όσα περισσότερα τόσο το καλύτερο. Αλλά όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ω πρόεδρος θα πρέπει και εγώ να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ας πω καταρχάς το εξής. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα αυτής της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για τέτοια ζητήματα στα πλαίσια του ΕΛΚΑ, πρέπει να σας πω ότι το ΕΛΚΑ σαφώς υποστηρίζει την αναφορά σας και σαφώς πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει κάθε τι το δυνατό για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βάσει όμως της συζήτηση αυτής, θα ήθελα να καταλήξω σε πέντε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα. Πρώτον, προφανώς η αναφορά αυτή θα μείνει ανοιχτή. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό ότι θα πρέπει να μην ανοιχτή αναφορά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το ζήτημα αυτό και να το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, να δούμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις. Το δεύτερο αίτημα το οποίο άκουσα μόλι τώρα ήταν να αποσταλεί μια διερευνητική αποστολή στην Ισπανία. Νομίζω ότι μπορούμε να καταγράψουμε και το αίτημα αυτό και να προωθήσουμε το αίτημα αυτό στην αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά στους συντονιστέ τη Επιτροπής μας. Αυτοί θα αποφασίσουν και θα συζητήσουν για την ενδεχόμενη αυτή διαρευνητική αποστολή. Να σα δώσω και τη δική μου προσωπική γνώμη. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι ισπανικές αρχές δεν δίνουν ενδεχομένω τη δέουσα σημασία στο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει πιο ηχηρά τα αιτήματά του και να ασκήσει κατά αυτόν τον τρόπο πίεση στι ισπανικέ αρχές προκειμένου να επιληφθούν με το δέοντα τρόπο με το ζήτημα αυτό. Τώρα, τρίτο συμπέρασμα. Η νέα Υπουργό Δικαιοσύνη είναι η πρώην εισαγγελέα κατά τη τρομοκρατία τη Ισπανία. Επομένω, θα τη αποστείλουμε και μια νέα επιστολή στην οποία θα λέμε ότι περιμένουμε πιο συγκεκριμένες πλέον απαντήσεις και πιο συγκεκριμένη ανάληψη δράσης πλέον από τις Ισπανικές Αρχές. Τέταρτο συμπέρασμα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έγγραφα, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε κτλ. θα πρέπει να πάνε στον Ισπανό συνήγορο του πολίτη, ο οποίος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης και θα μπορούσε να δει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε, αν θέλετε, και τη δική του εμπειρογνωμοσύνη για το ζήτημα αυτό. Αυτά πάνω κάτω θεωρώ μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο για αυτή την αναφορά. Νομίζω, διαισθάνομαι ότι υπάρχει μια συνένεση ανάμεσα στους συναδέλφους, έτσι δεν είναι. Και απευθυνόμενο στους αναφέροντες, το μόνο που μπορώ να πω είναι συνεχίστε τις δύσκολες αυτές προσπάθειές σας. Ξέρω ότι απαιτείται τεράστια ενέργεια για να επιληφθεί κανείς αυτού του ζητήματος, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε από κοινού να ασκούμε πίεση και προφανώς έχετε τη συμπαράσταση και την πλήρη συμπόνια των Ευρωπαίων Βουλευτών. Θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, όπως κάναμε και στο παρελθόν, έτσι θα κάνουμε και στο μέλλον. Δεν μπορούμε όμως εμείς να πάρουμε σε καμία περίπτωση τις τελικές αποφάσεις καθήλυνα αρμόδιοι είναι οι Ισπανικές αρχές και οι Ισπανικές δικαστικές αρχέ συγκεκριμένα. Αν είναι απόκειτο σε εμά θα είχαμε αποδώσει ήδη δικαιοσύνη, θεωρώ. Δυστυχώς όμως το ζήτημα αυτό εμπίπτει σαφώς στην αρμοδιότητα των Ισπανικών δικαστικών αρχών. Θα ήθελα να ξαναδώσω τώρα το λόγο για δύο λεπτά στους αναφέροντες. Ευχαριστώ. Ένα θέμα που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να διευκρινιστεί. Το βασικό ζήτημα είναι τα εγκλήματα που έκανε η ΕΤΑ και μόνο. Ε, η δεχθή, θηριώδη, κατά της ανθρωπότητας, όπως θέλετε πέστε τα. Αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Και δεν ζητούμε μόνο δικαιοσύνη, αλλά και δικαίωμα στην αλήθεια. Μίλα πιο αργά, λένε οι κυρίες εδώ, για, να, δείτε την ερμηνεία. Λέω, υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα, εκτός από τα ίδια τα εγκλήματα που λέγεται ατιμορρησία. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, για να μείνει πάρα πολύ σαφές σήμερα αυτό εδώ. Στις 25 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, κλείνουν 20 χρόνια από τη δολοφονία του Μανουέλ Θαμαρένιο. 20 χρόνια ατιμορρησίας. Η Ισπανία 20 χρόνια δεν την διερευνά αυτή την περίπτωση. Όπως και με τον Κάσο πριν από έξι μήνες, πρώτα σκότωσαν τον ένα και μετά τον άλλον. Πήγαμε στην Αργεντινή γιατί δεν το ψάχνει η ε, Ισπανία. Και στα πλαίσια της παγκόσμιας αρμοδιότητας το δέχτηκε η Αργεντινή και ε, ε, άνοιξε μια δικογραφία για Εδώ λοιπόν είναι η ατιμορρησία. Όταν η Αργεντινή όμω ζήτησε από την Ισπανία, γι' αυτό είναι το ψεύδος, όλα τα στοιχεία για να δει τι συνέβη, γιατί αποφάσισε να, διερευνήσει την περίπτωση Θαμαρένιο που δεν έψαχνε η Ισπανία και στα πλαίσια της παγκόσμια αρμοδιότητα καθολικής, τι απάντησε η Ισπανία, ότι οι περιπτώσει Κάσο και Θαμαρένιο έχουν εξηγνιαστεί και έχει επιβληθεί τιμωρία στους ε, ε, ενόχους. Αυτό είναι κατάφορο ψέμα και, και ξαδιάντροπο. Δεν γνωρίζουν κανένα όριο. Διότι είναι από μόνο του φοβερό και σοβαρό να έχει αφήσει ατιμόρυτους τους ε, δολοφόνους 20 χρόνια και πάνε τα θύματα, περνάνε τον Ατλαντικό, πηγαίνουν στον Buenos Aires, πληρώνουν δικηγόρο, ανοίγει η δικογραφία και η Ισπανία επίμονα αρνείται να το διερευνήσει. Δεν φτάνει ότι δεν το ερευνά, αλλά και άλλος δικαστής δεν έχει την πληροφόρηση και πάνε και λένε ψέματα στον ε, Αργεντινό ε, ανακριτή ότι δεν μπορείτε να το ψάξετε γιατί έχουν τιμωρηθεί ένοχοι. Ε, εδώ έχω επιστολές και θα σας τις δώσω από τις χείρε του Θαμαρένιο και του Κάσο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει δίνει. Είναι ψέματα αυτά δεν έχουν εξηχνιαστεί οι δολοφονίες Κάσο και Θαμαρένιο. Και χρειάστηκε να πάμε ε, χαρτί στην Αργεντινή από το συνήγορο του πολίτη από την Ισπανία που λέει ότι ψεύδονται οι Ισπανικέ αρχέ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να διερευνήσει αυτέ τι υποθέσει η Ισπανία και ψεύνεται. Ψεύδεται. Απαντάει γενικόλογα. Και έχουμε ε, ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ε, ε, ε, ο μηχανισμός Share Γιατί δεν το εφαρμόζει. αυτό που έχει γίνει στη Γερμανία, γιατί τους ξέρουν ποιοι είναι οι ηγέτες της ΕΤΑ. Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τολμάει, να ψεύδεται, να ψεύδεται και να εμποδίζει μια άλλη χώρα, ένα άλλο κράτος να διερευνήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί μια χώρα όπως η Ισπανία να πάει στην Αργεντινή και να πει ότι όχι, όχι, οι περιπτώσεις δολοφονίες Κάσο και Θωμαρένιο έχουν εξηχνιαστεί και αυτές οι χείρες που τις έχουν ξεχάσει 20 χρόνια να στέλνουν επιστολές και να εκλυπαρούν τον ανακριτή στην Αργεντινή να μην το βάλει στο αρχείο δεν είναι απόλυτη περιφρόνηση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των θυμάτων. Υπάρχει μεγαλύτερη ύβρις από αυτή, αφού έχουν αφήσει 20 χρόνια ατιμόρυτους τους δολοφόνους και τις έχουν πετάξει εκεί στην γωνία. Τι άλλο, προσπαθούν τώρα να εξαπατήσουν και έναν Αργεντινό δικαστή για να μην το διαρευνήσει. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα για κράτος μέλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλουμε να λάβετε υπόψη και είναι το νέο στοιχείο για το οποίο θα πρέπει να ρωτήσετε όταν πάτε στην Ισπανία. Και θα σας φέρουμε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Για να κλείσουμε, συνοψίζω, η αίτηση θα παραμείνει ανοιχτή. Η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή και θα προχωρήσουμε όπως σας περιέγραψα. Θα ζητήσουμε απάντηση από τον ε, Ισπανό του Πολίτη και θα επανέλθουμε συζητώντας το θέμα στην συνάντηση των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών. Θα απαιτεί συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε στην τελευταία αναφορά για σήμερα. Είναι η 665 του 2015, Γερμανού πολίτη, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του ερουλημένα της Φραγκφούρτης. Από όσο γνωρίζω δεν παρευρίσκεται ο αναφέρον. Εντάξει. Έχουμε όμως λάβει τα στοιχεία της αναφοράς του και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ανακρίβειες, ότι δεν είναι 100% αληθή αυτά που αναφέρονται στην αίτηση στην αναφορά, συγγνώμη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τη θέση της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γλυκά εγώ. Και νομίζω δεν θα χρειαστεί να μακρηγορήσω στο θέμα αυτό. Λάβαμε την αναφορά ε, του κυρίου αυτού και λέγεται σε αυτήν ότι ήταν απαράδεκτη να χρηματοδοτηθεί, απαράδεκτό να χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επέκταση του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης, γιατί αυτό, λέει, ε, σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ε, χρηματοδοτούν με τα χρήματά τους την αύξηση του θορύβου στην περιοχή. Γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την περιφερειακή ανάπτυξη στην, προηγούμενη, στην τρέχουσα μάλλον προγραμματική περίοδο δεν έχουμε κάποια χρηματοδότηση στον τομέα αυτό, αυτού του έργου. Υπάρχουν διάφορες προτεραιότητες αυτού του ταμείου που συμπεριλαμβάνουν τις μικρομερικές επιχειρήσεις, την καινοτομία, την έρευνα, αλλά όπως έχουμε ήδη απαντήσει στον αναφέροντα, στο πρόγραμμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία περίπτωση συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής δεν έχει υπάρξει καμιά τέτοια χρηματοδότηση μέχρι στιγμή και σε αυτό θα, θα μείνω. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστούμε κύριε Χέρν. Έχουμε αναλύσει και εμείς την αναφορά. Ε, φαίνεται ότι ίσως υπάρχει υπάρξει κάποια παρανόηση. Ίσως να μην ε, έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης, να μην γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί ο αναφέρον, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, κλείσουμε αυτή την αναφορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε τα θέματα της ημερησίας μας διάταξης. Θα κλείσουμε εδώ. Αύριο στις 9 θα έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών και στις 10.30 την τακτική μας συνεδρίαση. Ε, θα ξεκινήσουμε αύριο στις 10.30 με την ψηφοφορία. Καλό απόγευμα και γεια σας.